Ladies and gentlemen, may we start? Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμά μας με το σημείο υπαριθμών 30 και 8 ανταλλαγή απόψεων και δίνω το λόγο στην κυρία Λεγκρίπ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι σήμερα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε εν συντομία μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την πρόταση οδηγίας η οποία στοχεύει στην προστασία της γνώσεως και των εμπορικών ε, απορρίπτων. Γίνεται αυτή η συζήτηση μετά την πρώτη, όταν είχε παρουσιαστεί το σχέδιο κειμένου. Θέλω να υπενθυμίσω στο σύνολο των μελών μας ότι η αρχή μιας ε, ακρόασης έχει γίνει δεκτή ομόφωνα μεταξύ των μέλων της Επιτροπής μας και η εν λόγω ε, ακρόαση σε σχέση με τα λεγόμενα εμπορικά μυστικά θα γίνει τον Ιανουάριο με την ευκαιρία της συνεδρίασής μας του Ιανουαρίου. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δυστυχώς ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ούτε ξέρουμε καν τις πρακτικές λεπτομέρειες του γεγονότος αυτού αλλά τον Ιανουάριο παρόλα αυτά θα λάβει χώρα αυτή η ακρόαση σε μια κομβική στιγμή που θα σας επιτρέψει να ακούσετε τις απόψεις των διαφόρων εμπλεκομένων ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη γνώση μας για τα θέματα αυτά και να έχουμε μια καλύτερη προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης που έχω την τιμή ή υποφαινομένη να παρουσιάσω ενώπιον της Επιτροπής σας. Επομένω με την ακρόαση αυτή κάπω θα καθυστερήσει το σχέδιο χρονοδιαγράμματος που σα είχα παρουσιάσει την προηγούμενη φορά. Το σχέδιο έκθεσης που με μεγάλη τιμή θα σας παρουσιάσω θα κατατεθεί κατόπιν της ακροάσεως τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου Θεού θέλοντος θα συζητήσουμε στη συνεδρίασή μας που προβλέπεται για τις αρχές Φεβρουαρίου και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εκτίληξη των εργασιών μας μεταξύ του, της εισηγήτριας και των σκιωδών με τρόπο καρποφόρο ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή στην συνεδρίασή μας στα μέσα Απριλίου. Βρισκόμαστε ακόμα σε επίπεδο μελέτης του κειμένου που παρουσίασε η Επιτροπή πληροφορούμεθα σε σχέση με τα θέματα αυτά, μελετούμε τις συγκριτικές έρευνες που έχουν γίνει, εξετάζουμε το κείμενο το οποίο ενεκρίθη από το Συμβούλιο, διότι το Συμβούλιο έχει ήδη την ευκαιρία να εκφράσει γνώμη για το κείμενο αυτό αρκετά ταχαίως και προχωρεί με διαβουλεύσεις μεταξύ εμπλεκομένων, επιχειρηματιών, ε, λομπιστών, εργαζομένων, διανοουμένων, την Ένωση των Ευρωπαίων Νόμομαθών Επιχειρήσεων, που έχουν πολλά πράγματα να πούνε. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτή τη βασική διαπίστωση και θέλω να συμμεριστώ μαζί σας ορισμένα στοιχεία τις σκέψεις μου και ορισμένα σχόλια και παρατηρήσεις που ήλξα από την διαβούλευση η οποία έχει λάβει η χώρα και η οποία θα ακολουθηθεί από άλλες διαβουλεύσεις. Πρώτο σημείο μου φαίνεται κεφαλαιόδες να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της οδηγίας. Πιστεύω ότι ως έχει αυτή τη στιγμή η οδηγία αυτή η οποία βρίσκεται στο τραπέζι μας, οι επιχειρήσεις μπορεί να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα σε σχέση με την αποτελεσματική ε, προστασία των εμπορικού χαρακτήρα απορρίτων πληροφοριών τους. Νομίζω ότι μέσα στο σχέδιο της οδηγίας ως έχει υπάρχουν κάποιες διατάξεις οι οποίες δεν έχουν επαρκές βάρος και ακρίβεια και θα ήταν χρήσιμο να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ορισμένα αποτρεπτικά στοιχεία που θα εμποδίσουν τις παραβιάσεις και να <clears throat> μειώσουμε τις ε, πιέσεις και τους περιορισμούς διαδικαστικού χαρακτήρα που μπορεί να εμποδίζουν τις επιχειρήσεις όταν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Τα στοιχεία απόδειξης, παραδείγματος τα αποδεικτικά στοιχεία, όπως λέει το άρθρο 3 που πρέπει να παρουσιαστούν από τους προσφεύγοντας ή το διάστημα παραγραφής όπως αναφέρεται στο σημείο 7. Δεύτερη παρατήρηση θέλω να αναφερθώ στο σημείο 8 για την προστασία του εμπορικού απορρίτου σε νομικές, σε δικαστικές διαδικασίες. Αυτό είναι κομβικό για την αποτελεσματικότητα αυτής της οδηγίας και το Συμβούλιο σκέφτηκε πολύ για το άρθρο 8 και πάλι <clears throat> έχει προταθεί ένα καινοτόμο στοιχείο στην περίπτωση αυτή το οποίο όμως θα πρέπει να διευκρινιστεί καλύτερα το θέμα της αντιπροσωπευτικότητας των ε, ε, εμπλεκομένων μερών για την πρόσβασή τους σε εμπιστευτικά έγγραφα και επίσης η διαδικασία για την διαμειουργία προστασίας του απορρίτου και αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο. Μια ακόμα παρατήρηση θα ήθελα να σας αναφέρω ότι η προσοχή μας εστιάστηκε πολλές φορές στο θέμα της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που δίδονται στις ε, αρχές που κατακυρώνουν ένα δημόσιο διαγωνισμό. Μερικές φορές οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να σεβαστούν και είναι πολύ αυστηρή αυτή η διαδικασία, ότι μπορούν να σεβαστούν στη συγγραφή υποχρεώσεων που ουσιαστικά σημαίνει ότι πρέπει να δώσουν στοιχεία που είναι εμπορικά απόρριτα. <clears throat> Αυτό σημαίνει ότι βαραίνει μια σημαντική ευθύνη την κατακυρώνουσα αρχή, τι δημόσιε αρχές οι οποίε είναι υπεύθυνε για του δημόσιους διαγωνισμούς, έχουν λοιπόν μια σημαντική ευθύνη και την οποία δεν πρέπει να παραβιάσουν κάνοντα μια καταχρηστική χρήση των πληροφοριών που αποκτούν κατά τη διάρκεια του δημόσιου διαγωνισμού, γιατί αυτό ήταν σε βάρο του συμφέροντος των ε, διαγωνιζομένων. Οι δημόσιες αρχές όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το εξής, ότι θα είναι απαραίτητο να βρούμε τα απαραίτητα εργαλεία ώστε ούτως πίν να καταγράψουμε αυτή την ευθύνη των δημοσίων αρχών και να την ενσωματώσουμε στην οδηγία. Δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω πρόοδο. Τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω σε αυτό το στάδιο της συζήτησης, κάτι το οποίο μου φαίνεται ένα δύσκολο ακαθόδες θέμα και το οποίο αναφέρθηκε πολλές φορές στις ε, συζητήσεις που έκανα μέσα στη διαβούλευση, είναι το θέμα των συμβατικών σχέσεων μεταξύ ενός εργαζομένου, ενός εργοδότη, και των ε, ε, εργαζομένων, των μισθωτών του. Οι πληροφορίες λοιπόν που αποκτούν οι μισθωτοί καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης του επαγγελματός τους, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβαση αυτής, κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες όταν εκπνεύσει αυτό το συμβόλαιο. Η προστασία λοιπόν των επιχείρησεων εναντίον μιας επιθετικής στάσης που μπορούν να κρατήσουν κάποιοι εργαζόμενοι πρέπει να τύχει εγγύησης. Το να μην υπάρχει, ε, να μην δουλέψουν για τους ανταγωνιστές τους αυτοί όπως υπάρχει σε ορισμένα συμβόλαια, αυτό μερικές φορές είναι απόλυτα δικαιολογημένο, αλλά υπάρχει εδώ ένα λεπτό θέμα, η απόλυτη προάσπιση του εμπορικού απορρίτου σε αυτήν την περίπτωση, που είναι υπερβολικά, θα μπορούσε η αυστηρή, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταχρηστικές ενέργειες, θα μπορούσε σε ορισμένε περιπτώσεις να περιορίσει και την κινητικότητα και την ελευθερία κίνησης των εργαζομένων μετά το τέλος του συμβολέου τους. <clears throat> αυτά λοιπόν πρέπει να τα προσέξουμε, το τονίζει και η οδηγία ότι είναι λεπτά τα θέματα αυτά, είναι απαραίτητο όμως να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο, χωρίς να βγούμε από τα χωράφια αρμοδιότητάς μας, αλλά και να μην φτιάξουμε διατάξεις οι οποίες βγαίνουν και έξω από την ευρωπαϊκή αρμοδιότητα και δεν έχουν νομική βάση, αλλά για μια ακόμα φορά είναι απαραίτητο να καταπιαστούμε με το θέμα αυτό και να λάβουμε υπόψη τις απόψεις των εμπλεκομένων. Αυτά λοιπόν κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας τα πω εν συντομία να σας παρουσιάσω ορισμένες πτυχές του προβλήματος αυτού. Πιστεύω ότι στα σημεία αυτά θα μπορούσαμε να έχουμε μία συζήτηση με την ε, ευκαιρία της ακρόασης του Ιανουαρίου. Θα ήθελα να μπορέσω να συζητήσω με τους σκιώδεις συζητητές από όλες τις πολιτικές ομάδες, ώστε να αποδηθούμε σε μια κοινή συζήτηση και ένα κοινό προβληματισμό. Είναι η πρόθεσή μου στις επόμενες εβδομάδες να συναντήσω όλους τους τους συζητητές και να τους προτείνω μια πρώτη συνάντηση εργασίας, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο σημείο αυτό με τρόπο ουσιαστικό τις εργασίες μας. Και κλείνω, λέγον κύριε Πρόεδρε, υπενθυμίζουν για μια ακόμα φορά πόσο χρήσιμο είναι να έχουμε ένα τέτοιο σχέδιο οδηγίας μέσα στο τωρινό οικονομικό πλαίσιο. Το κομβικό θέμα εδώ νομίζω ότι είναι αυτό της εμπιστοσύνης, το να μπορέσουμε να έχουμε ένα νομοθετικό μέτρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο έχει εναρμονισμένο χαρακτήρα και το οποίο ξεπερνά τον τωρινό κατακαιρματισμό του δικαίου για τα θέματα αυτά. Αυτό θα εξυπηρετήσει ιδιαίτερα την εσωτερική αγορά σε ό,τι αφορά την προστασία των ε, εμπιστευτικών εμπορικών πληροφοριών και της τεχνογνωσίας που είναι βέβαια στην καρδιά του ρόλου μιας επιχείρησης και θα μας επιτρέψει να έχουμε μια περαιτέρα εδραίωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς αλλά και να δημιουργήσουμε και ένα υπόβαθρο ασφάλειας, προστασίας και εμπιστοσύνης που είναι απαράγραπτο για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε οικονομικά τις επιχειρήσεις μας την ίδια αυτή Ευρωπαϊκή Ήπειρο και επίσης να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ικανότητα του καινοτομήν και του ανταγωνίζεστε. Λοιπόν, το σύνθημά μας είναι εμπιστοσύνη, όχι να φτιάξουμε πετάσματα και φράγματα, αλλά να δημιουργήσουμε το έφορο υπόβαθρο εμπιστοσύνη για να εξασφαλίσουμε περισσότερη καινοτομία και ανταγωνιστικότητα που χρειαζόμαστε τόσο πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, madam. Now the... Σας ευχαριστώ. Απόψη σχόλια. Ευχαριστώ. Δύο λόγια. Πρώτον, Ευχαριστώ την κυρία Λεγκρίπ για την αντικειμενικότητα της εκθέσεως. Σημαντικό αυτό. Το ζήτημα της δημοσίας τάξης δηλαδή και η κινδύνη για το επιχειρηματικό απόρριτο επίσης αθέμητο συνταγωνισμό κλπ. που θα τεθεί αύριο και θα αποτελεί ένα από του κινδύνου. Έναν από τους κινδύνους. Εγώ θα ήθελα τώρα μόνο στο όνομα του Ζουλιά Ρεντάκ που δεν είναι παρόν και που παρακολουθεί το θέμα από πλευράς των Πρασίνων να εφιστήσουν την προσοχή και της Κομισιόν και της κ. Λεγκρίπ στον ευρύ χαρακτήρα του επιχειρηματικού απορρίτου. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παράδοξο. Έχω ξαναμιλήσει σε ένα ενδιαφέρον ραντεβού εργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε ένα γενικό όρο και μερικές εξαιρέσεις. Αυτό το ζήτημα το κοινωνικό είναι πολύ περιορισμένο. Το ζήτημα είναι ποιο είναι το προστατευταίο αγαθό. Εκεί όπου δεν μπορούν τα πράγματα αυτά να μπουν μέσα σε πολύ περίπλοκους ε, νομικούς μηχανισμούς. Τι ακριβώς είναι λοιπόν το επιχειρηματικό απόρριτο, ποιο είναι το συμφέρον που νομιμοποιείται για να προστατευτεί δεν είναι δυνατόν δηλαδή να αρκεστούμε μοναχά σε μια περιγραφή ενό γενικού όρου. Διευκρίνηση λοιπόν του επιχειρηματικού απορρίτου, διευκρίνηση του νόμιμου συμφέροντος που αξίζει προστασίας. Κύριε Κοφεράτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Λεγκρίπ και θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις για την εργασία που ξεκίνησε και που θα κάνουμε από κοινού. Η πρώτη παρατηρήση είναι γενικού χαρακτήρα. Εμείς πρέπει, επειδή αυτό μας ζητάει η Κομισιόν, να στοχεύσουμε σε μια υπεράσπιση των πληροφοριών που μπορούν να ε, παρουσιάζουν μια προστιθέμενη αξία λόγω της δραστηριότητας και του αντικειμένου. Ε, αυτό είναι δυνατόν μέσα από αυτή εδώ την ε, πρόταση. Εγώ πιστεύω πως είναι σκόπεμο η... τα νομοθετήματα να εγγυώνται τέτοιου είδους πληροφορίες. Ωστόσο πρέπει να προσέξουμε πολύ ώστε να βρούμε μια σωστή ισορροπία προς το κοινό συμφέρον των επιχειρήσεων, έτσι ώστε δηλαδή να μην καταστεί τόσο άκαμπτη η προστασία σε βαθμό που να εμποδίσει οι φυσιολογικές πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την καινοτομία και τη γνώση και ίσως και να ε, παροτρύνουν τον θεμητό ανταγωνισμό να περιορίζονται από αυτόν το νομοθέτημα. Είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να το πει κανείς, αλλά είναι πιο δύσκολο να το εντοπίσει κανείς, ακριβώς γιατί πρέπει να βρεθεί, όπως είπα, η κατάλληλη ισορροπία. Δεν είναι κάτι το οποίο ήδη είναι εδρεωμένο από την πρακτική και άρα θα πρέπει να το εφεύρουμε και να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας. Ε, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να είμαστε σαφείς όσον αφορά το χαρακτήρα του νομοθετήματος αυτού. Δεν θέλουμε να ορίσουμε ένα νέο είδος ε, διπλώματος ευρεσιτεχνία χαμηλού επίπεδου από αυτό με το οποίο ήδη έχουμε ασχοληθεί αν υπάρχουν θέματα που αφορούν ε, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ε, θα πρέπει να επιληθούν μέσω του αντίστοιχου νομοθετήματος, όχι μέσω αυτού εδώ. Ε, εδώ ο στόχος είναι αυτό που θύμισε επανειλημμένα η συνάδελφος, ότι δηλαδή χρειάζεται να υπάρχουν πληροφορίες, μάλλον να μην γίνεται χρήση άσκοπη των πληροφοριών που αφορούν το εσωτερικά την κάθε επιχείρηση. Γι' αυτό θα απαιτηθεί πολύ προσοχή όσον αφορά τον ορισμό τον ακριβή του τι ακριβώς εννοούμε μέσω της φράσης αυτής που λέμε παράνομη απόκτηση. Γι' αυτό για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως, ότι δηλαδή ότι υπάρχει μια πολύ λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις γνώσεις, κυκλοφορία γνώσεων από τη μια πλευρά και προστασία των στοιχείων που αντικειμενικά αποτελούν απροστεθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις. Και το λέω και επιμένω σε αυτή την πτυχή, διότι είναι σημαντική ε, όσον αφορά την τρίτη παρατηρήση που θέλω να κάνω, το είπε η συνάδελφος και συμφωνώ μαζί της, ότι δηλαδή πρέπει να αφιερώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες τις οποίες επεξεργάζονται οι εργαζόμενοι, ειδικά οι εργαζόμενοι ψηλά ειστάμενοι στην άσκηση των καθηκόντων τους. Για αυτούς είναι φυσιολογική διαχείριση πληροφοριών που είναι τμήμα της συστήματος της επιχείρησης, αλλά είναι και φυσικό οι πληροφορίες αυτές σε μεγάλο βαθμό να προκύπτουν χάρη στη δική τους δημιουργική ικανότητα. Ταυτόχρονα λοιπόν αποτελούν προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση, αλλά και ε, θεμέλιο της επαγγελματικότητάς τους. Όπως γνωρίζετε, συμβαίνει συχνά εργαζόμενοι ψηλού επίπεδου να αφήνουν μια επιχείρηση για να, αναλάβουν, να κάνουν μια δική τους ατομική συλλογική δραστηριότητα. Και αυτό το κάνουν επί τη βάση της εμπειρίας τους που έχει οριμάσει, για να γνωρίζουν ότι έχουν αποκτήσει αυτές τις γνώσεις. Και εδώ δεν είναι εύκολη η διάκριση. Θα πρέπει πολύ προσεκτικά να ε, δουλέψουμε. Και, αλλά να προσέξουμε να μην εμποδίσουμε την πνευματική ανάπτυξη του εργαζόμενου που ασχολείται με την έρευνα και που ταυτόχρονα είναι χρήσιμη η γνώση που αναπτύσσει για την ίδια την εταιρεία του, αλλά μπορεί να αποτελέσει και δική το δικό του κληροδότημα, δική του, την ίδια δραστηριότητα σε έναν άλλο χώρο. Είτε είναι αυτό μια ατομική δική του επιχείρηση, είτε είναι άλλη συλλογική εργασία. Για αυτή λοιπόν την ε, πτυχή των εργαζομένων που είναι οι πιο υψηλά εκπαιδευμένη για αυτά τα θέματα, ε, θα πρέπει να προσέξουμε να φροντίσουμε να προστατεύσουμε το παραγωγικό τμήμα ε, χωρίς να αποθαρρύνουμε τη διάδοση του πολιτισμού, να εμποδίσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό και την άσκοπη χρήση των πληροφοριών, αλλά όχι την ε, πολιτιστική πνευματική ανάπτυξη που περνά πάντα από τη γνώση και την πράξη μέσα σε ίδια δραστηριότητα και τη δική μας συμπεριλαμβανομένη. Και οι βουλευτές έχουν πληροφορίε πολλές φορές που δεν ε, υπόκειται σε κανένα είδο έλεγχο, αλλά που συχνά ε, άλλες φορές χρησιμοποιούνται σε άλλες δραστηριότητε. Ευνοούμε λοιπόν σημαντικές δραστηριότητε ώστε να χωρίς να εμποδίσουμε την εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιάς, παρακαλώ να είστε σύντομο όμως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Το 2014 η Financial Times δημοσίευσε ένα κανόνα, ένα κατάλογο των 10 πρώτων εταιριών σε ό,τι αφορά την ε, αξία της επιχείρησής τους. Γιατί είναι οι περισσότερες αμερικανικές. Γιατί υπάρχει ένας νόμος για το εμπορικό απόρριτο που έχει εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει ενημερωθεί έκτοτε και δίδει τη δυνατότητα να υπάρχει ενημερωμένη διαδικασία για τα εμπορικά απόρριτα εταιρεών των ΗΠΑ που εργάζονται σε διάφορα μέρη. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλέ εταιρείε στι ΗΠΑ οι οποίε χρησιμοποιούν αυτό το εμπορικό απόρριτο για να έχουν μια ανταγωνιστική θέση. 75% των ε, απαντώντας σε μια έρευνα είπαν ότι το εμπορικό απόρριτο είναι κεφαλαιόδε για να εξασφαλίσει κανείς την ανταγωνιστικότητα. Παρόλα αυτά, στα πλαίσια του, της προστασίας ε, του εμπορικού απορρίτου υπάρχει έλλειψη εναρμόνισης στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι λοιπόν ε, ιδιαίτερα ε, επίκαιρη η πρόταση της Κομισιόν, μάλλον έρχεται και κατόπιν εορτής κατά κάποιο τρόπο. Πρέπει να υπάρξει μια αντιμετώπιση αντίστοιχη με αυτή των ευρεσιτεχνιών, να είναι ομοιόμορφη και νομίζω ότι μια τέτοια αριθμίση θα είναι πάρα πολύ θετική για τις επιχειρήσεις, θα βοηθήσει να έχουν ασφάλεια δικαίου σε σχέση με τις συναλλαγές τους. Πιστεύω ότι αυτή η πρόταση οδηγίας θα διευκολύνει τα μάλα το έργο και των εθνικών δικαστηρίων σε περίπτωση ε, μη νόμιμης απόκτησης και χρήσης εμπορικών απορρίτων. Θα διευκολύνει επίσης και τη διαδικασία αποζημίωσης των θυμάτων. Εγώ υποστηρίζω την πρόταση του Συμβουλίου για μια πιο εξισορροπημένη προσέγγιση στην προστασία των εμπορικών ε, μυστικών και του δικαιώματος μιας δίκαιας δίκης. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι είναι μακρά η περίοδος παραγραφής για να έχουν μεγαλύτερη προστασία αυτών των απορρίτων. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ροζιέρ. Σας ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη σαφή της παρουσίαση των διακυβευμένων σε αυτή την οδηγία. Απλώς μερικές ε, σκέψεις που ήθελα να αναφέρω. Μιλάμε για ένα καθεστώς προστασίας του εμπορικού απορρίτου που φυσικά μπορεί να έχει αχανή χαρακτήρα λόγω της φύσης του. Ίσως η ακρόαση που θα κάνουμε θα διευκρινίσει καλύτερα τα θέματα αυτά, αλλά λόγω της έκταση αυτού του θέματος να έχουμε την προστασία των εμπορικών μυστικών, όταν έχουμε και ένα καθεστώς για την πνευματική ιδιοκτησία που προστατεύει τις πληροφορίες στα πλαίσια μια επιχείρησης εφόσον γίνουν δημόσιες, Βλέπουμε εδώ ότι με ένα καθεστώς προστασίας το οποίο φαίνεται ιδιαίτερα γενικό σήμερα και αρκετά ευρύ, για αυτό το σύστημα δεν μπορούμε, όπως στην περίπτωση της πνευματικής ιδιοκτησίας, να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει και το δημόσιο των πληροφοριών αυτών. Τόσο γενικός χαρακτήρας του ορισμού του εμπορικού απορρίτου στο άρθρο 4 που αναφέρει τι είναι θεμητό σε ό,τι αφορά την απόκτηση εμπορικών απορρίτων, νομίζω ότι περιλαμβάνει υπερβολικούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά την ε, διαβίβαση αυτών των απορρίτων και πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης εξασφάλισης ε, ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά επίσης και να προστατεύει τους άλλους εμπλεκομένους όπως είναι οι εργαζόμενοι, η κοινωνία των πολιτών οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να έχουν κάποιες από αυτές τις πληροφορίες που αποτελούν ε, εμπιστευτικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η τελευταία <clears throat> παρέμβαση. Όχι, συγγνώμη και εσείς, η κυρία Γκούτε Λάντ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και την εισηγήτρια θα ευχαριστήσω για την πολύ καλή παρουσίασή της. Κατανοώ την ε, πρόθεση και την καλή πρόθεση μάλλον αυτή τη πρόταση, θέλω να υπογραμμίσω κάτι άλλο. Τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πρώτα απ' όλα θέλω να αναφέρω την ανησυχία μου σε σχέση με τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το θέμα της εκπροσώπησης και της πληροφόρησης των εργαζομένων. Ιδιαίτερα σε πολλά κράτη-μέλη που περιλαμβάνουν και το δικό μου τη Σουηδία, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα έχουν το δικαίωμα να έχουν ένα εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους με ουσιαστικό τρόπο. Τι αντίκτυπο όμως θα μπορούσε να έχει αυτή η πρόταση σε σχέση με το δικαίωμα πληροφόρησης και εκπροσώψης των εργαζομένων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, σε κάποια κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και τη Σουηδία, η ρύθμιση για τα θέματα αυτά επαφίεται στους κοινωνικούς εταίρους. Μέχρι στιγμής αυτό έχει λειτουργήσει πολύ καλά ήταν ένας καλός τρόπος να έχουμε λύσεις οι οποίες ήταν επωφελείς μέσω συλλογικών συμφωνιών. Έχει λάβει υπόψη η Κομισιόν τα διατύπωση στην πρόταση αυτή τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεάσει τις χώρες όπου λειτουργούν αυτές οι συλλογικές συμβάσεις και συμφωνίες. Τι θα συμβεί με τις λύσεις οι οποίες επιτυγχάνονται μέσω του κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμφωνιών και όχι με νομική ρύθμιση. Αυτό θα έχει μια άμεση και έντονη επίδραση σε χώρες όπως η δική μου. Τρίτον, μια γενικότερη ανησυχία. Αν υπάρχουν μέτρα τα οποία προχωρούν πολύ μακριά στον τομέα αυτό, μπορεί με τον τρόπο αυτό να περιοριστεί η ικανότητα των εργαζομένων να αντλούν από την προηγούμενη εργασιακή τους εμπειρία και να χρησιμοποιούν τη γνώση που έχουν αποκτήσει όταν πηγαίνουν σε μια άλλη θέση εργασίας μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Φοβάμαι ότι με τον τρόπο αυτό θα υποχρεώνονται οι εργαζόμενοι να παραμένουν στην αρχική τους επιχείρηση και θα μειώσει και την κινητικότητα. Έχει σκεφτεί για αυτά τα θέματα η Κομισιόν. Αυτό είναι η ανησυχία που θέλω να εκφράσω. Ε, ε, Κυρία Λεγκρίπ, θέλει να κάνει κάποια σχόλια, όχι. Εντάξει. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο μάλλον. Και όλα αυτά τα θέματα που έχουν διατυπωθεί, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να τύχουν απαντήσεις. Ούτως κλείνουμε το σημείο αυτό και περνάμε στο σημείο 39 ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την σύναψη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ε, συνθήκης του Μαρακές για να διευκολυνθεί η δυνατότητα εργασίας ανθρώπων που είναι τυφλοί ή έχουν κάποια άλλη ανυπηρία, αναπηρία. Ο κύριος Αντεσόνα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά την ε, Μαρία Μάρτιν Φράτ από την ε, Κομισιόν. Ελπίζω να έχει ήδη φτάσει. Θα έλεγα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ευτυχές που η Κομισιόν υπέγραψε τη συνθήκη και αυτή η μεταρρύθμιση είναι κάτι που οι πράσινοι ήθελαν εδώ και πολύ καιρό και έχουν αγωνιστεί γι' αυτό. Θα ήθελα να καλέσω την εκπρόσωπο της Κομισιόν λοιπόν να μας πει περισσότερα για την πρόταση καθώς και για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. So the floor would be to, uh, Μάλιστα, να δώσουμε λοιπόν το λόγο στην Κομισιόν, στην κυρία Πράτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ θετικά τα νέα για την Κομισιόν που μπορούμε να σας πούμε στις 31 Οκτωβρίου η Κομισιόν υιοθέτησε την πρόταση για, πρόταση, ε, για απόφαση μάλλον του Συμβουλίου για τροποποίηση της συνθήκης του Μαρακές. Να σας ε, ενημερώσω σύντομα γιατί ξέρω πως ε, είσαστε πολύ εξοικειωμένοι με το θέμα αλλά να σας πω το ιστορικό, η συνθήκη του Μαρακές ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό ε, Πνευματικών Δικαιωμάτων. Η Κομισιόν διπλωματεύτηκε εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της και η συνθήκη αυτή υιοθετήθηκε σε διπλωματική διάσκεψη τον Ιούνιο του 2013. Στη συνέχεια ε, πρέπει πάντοτε να γίνουν δύο βήματα, υπογραφή της συνθήκης και μετά επικύρωση αυτής. Η, πρόταση, η Κομισιόν μάλλον σύντομα μετά την διπλωματική διάσκεψη και την ολοκλήρωση αυτής ε, της συνθήκης υποβάλαμε σύντομα την πρόταση για την υπογραφή της συνθήκης το Δεκέμβριο του 2013 και τελικά υιοθετήθηκε και υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2014. Και τώρα έχουμε θέσει στο τραπέζι του Συμβουλίου την πρόταση αυτή προς ε, επικύρωση. Φυσικά πρόκειται για μια πρόταση που θα έρθει και σε εσά, διότι το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να δώσει την σύμφωνη, τη συγκατάθεσή του πριν υιοθετηθεί η απόφαση. Βασικά δηλαδή αυτό που ζητάμε από το Κοινοβούλιο είναι πολύ απλό να να επιτρέψει την επικύρωση της ηθίκης ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση για τα άτομα που είναι, που έχουν, που είναι τυφλοί ή έχουν δυσκολία στην όραση ή έχουν κάποια διαφορετική ε, άλλη μάλλον αναπηρία. Έτσι, μετά από την επικύρωση της συνθήκης ε, όπου απαιτούνται 20, 20 επικυρώσεις στην αρχή να ισχύει για την ώρα μόνο τρεις χώρες έχουν επικυρώσει Τη συνθήκη είναι η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ελ Σαλβαδόρ. Αλλά ε, στο σύνολο είναι 80 οι χώρες που έχουν υπογράψει τις φόρες. Αυτό σημαίνει στην ουσία δέσμευση για επικύρωση. Αυτή είναι η κατάσταση προόδου. Η πρώτη συζήτηση με το Συμβούλιο θα γίνει Πρώτα στο επίπεδο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου, όπου προβλέπεται συνεδρία στις 24 του τρέχοντος μήνα. Στη συνέχεια έχουμε μια πρώτη συζήτηση. Δεν είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε νωρίτερα, γιατί όπως είπα η απόφαση ε, να εκρήθη πριν από τρεις εβδομάδες. Μετά από την πρώτη συζήτηση λοιπόν θα είμαστε σε θέση να σας υποδείξουμε πόσο γρήγορα πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει το θέμα και κατά πόσο υπάρχουν ειδικά προβλήματα που θα τα αναφέρει το Συμβούλιο. Αυτά μπορώ να σας πω για την ώρα, αλλά φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω οποιαδήποτε άλλη ερώτηση έχετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής θέλει να ξαναπάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο περαιτέρω ερωτήσεις. Η πρώτη είναι να μας πείτε κάπως περισσότερα πράγματα όσον αφορά την άποψη της Κομισιόν για το θέμα των αρμοδιοτήτων όσον αφορά την επικύρωση της συνθήκης του Μαρακές. Το δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξής. Το Κοινοβούλιο, όπως κατάλαβα, επισήμως δεν έχει λάβει το αίτημα το επίσημο αίτημα για να δώσει τη συγκατάθεσή του. Μπορείτε να μας ευκρινίσετε αυτό το θέμα παρακαλώ. Κυρία Μάρτιν Πράτ. Σας ευχαριστώ. Πρώτη ερώτηση. Αρμοδιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το αντικείμενο που καλύπτει η συνθήκη είναι αποκριστικής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό για μας είναι σαφές. Δεν είναι βέβαια και καινούργια συζήτηση αυτή. Νομίζω μάλιστα σήμερα το πρωί συζητούσατε την Conditional Access Convention του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν κάνει τις ίδιες συζητήσεις. Αποκλειστική ή κοινή αρμοδιότητα, μεικτή αρμοδιότητα λόγω της υφισταμένης νομοθεσίας αλλά και διότι γίνονται και ανταλλαγές με τρίτες χώρες. Το αντικείμενο λοιπόν τη συνθήκη του Μαρακές κατά τη γνώμη μας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ένωση. Σε ό,τι αφορά τώρα την επίσημη διαβίβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έγγραφο, η πρόταση δηλαδή αποφάσεως του Συμβουλίου είναι δημόσιο κτήμα και υπάρχει και, στο, και στην ιστοσελίδα Eurolex. Θεωρούμε ότι θα διαβιβαστεί επισήμως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο όταν θα έχει διεξαχθεί συζήτηση στο Συμβούλιο Υπουργών και τη στιγμή εκείνη πριν να λάβει θέση, μάλλον έχοντας λάβει θέση το Συμβούλιο, αλλά πριν να λάβει οριστικά απόφαση, επισήμως απόφαση, διαβιβάζει το κείμενο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι βεβαία ωστόσο ότι μπορούν να επιβεβαιώσουν οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου την διαδοχική σειρά αυτή των γεγονότων. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς έτσι λειτουργεί. Δεν είναι πάντως διαβάθμισμένο εγγραφό. Είναι δημόσιο και μπορεί ο καθένας να το συμβουλευτεί. Σας ευχαριστώ για την πολύ σαφή απάντησή σας. Ο Πρόεδρος. Καλά λοιπόν, έχουμε σχόλια από άλλα μέλη. Δεν βλέπω κανείς να σηκώνει το χέρι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι για σήμερα κλείνουμε τη συζήτηση του θέματος αυτού και μπορούμε να περάσουμε στο θέμα υπαριθμών 4 που το θέμα από μόνο του εξηγεί το πολυπληθές του ακροατηρίου μας. Καλώς ορίσατε όλες και όλοι λοιπόν στην ακρόαση για την μελλοντική εξέλιξη του copyright στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επιθυμώ να καλωσορίσω ιδίως την συμπρόεδρό μας Σίλβια Κώστα, πρόεδρο της ε, Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων που συνδιοργανώνει μαζί μας την ακρόαση. Η σημερινή ακρόαση είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, ιδίως από τότε που ο Jean-Claude Juncker, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοίνωσε ότι η μεταρρύθμιση του copyright στην ψηφιακή κοινωνία και οικονομία είναι μεταξύ των πρώτων 10 προτεραιοτήτων της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι όμως σημαντικό το θέμα σήμερα εξάλλου και για δύο άλλους λόγους. Αφενός την ανανεούμενη έμφαση που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην βελτίωση της νομοθεσίας και στο σχετικό θεματολόγιο, αλλά και λόγω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την συμφωνία με τις ΗΠΑ, την TTIP, που θέτει θέματα και ρυθμιστικά, αλλά και ε, πνευματικών διανοητικών ε, δικαιωμάτων σημειώστε ότι η σημερινή ακρόαση δεν θα ρίξει μόνο φως σε ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το copyright σήμερα στην Ευρώπη, θα αποτελέσει και το εφαλτήριο για δύο project που θα συνδιαμορφώσουν τις δραστηριότητες της Επιτροπής μας τα επόμενα χρόνια. Πρώτον, η Επιτροπή μας αποφάσισε να δημιουργήσει νέα ομάδα εργασίας για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησία και τη σχετική μεταρρύθμιση και μόλις χθε οι συντονιστέ τη Επιτροπής μας αποφάσισαν να ορίσουν τον Ζαν Μαρί Καβαντά, αντιπρόεδρο, ως συντονιστή αυτή τη ομάδα εργασίας, η οποία ομάδα εργασίας θα αποτελείται από ένα μέλος από κάθε μια πολιτική ομάδα που εκπροσωπείται στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και επίσης από την Επιτροπή Πολιτιστικών ε, Ενίας Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών και Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας. Θα συναντώνται άπαξ του μηνός, θα προσκαλούν και ειδικού για να συζητούν θέματα copyright σήμερα στην Ευρώπη. Δεύτερο, εκ με αυτή την ομάδα εργασίας η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία better regulation που έχει στη διάθεσή της, ώστε να προπορεύεται της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο προπαρασκευαστικό και αναλυτικό έργο της για την σύνταξη προτάσεων για το copyright. Ιδίως η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα συντάξει έκθεση εφαρμογής για την οδηγία για την αρμόνιση ορισμένων πτυχών του copyright και σχετικών δικαιωμάτων στην κοινωνία των πληροφοριών. Και ως πρώτο βήμα η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία μελετών του Ευρωκοινοβουλίου να προβεί σε μελέτη αντικτύπου ex post για την οδηγία, τα αποτελέσματα της οποίας θα, ε, θα συζητηθούν σε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς αλλά και με μελέτες εξάντε εκ των προτέρων που θα διεξαχθούν όλες αυτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραλλήλου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια το σχέδιο είναι πολύ φιλόδοξο και έχουμε πολύ σημαντικές ελπίδες ότι θα προκύψει έργο από αυτές τις προσπάθειες και βεβαίως είναι και συναρπαστική η εξέλιξη αυτή. Είναι σήμερα μια θαυμάσια μέρα για το copyright στην Ευρώπη. Με μεγάλη ανυπομονησία αναμένω τις παρεμβάσεις των ειδικών για τη συζήτηση για το μέλλον του copyright στην Ευρώπη. Πρώτα όμως θέλω να δώσω το λόγο στην συμπρόεδρό μου για να προβεί και αυτή σε εναρκτήριες ε, παρατηρήσεις για το θέμα. Δίνω το λόγο στην κυρία Σίλβια Κώστα που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτιστικών. Σας ευχαριστώ όλους, αλλά θα προτιμώ να μιλήσω στα Ιταλικά. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον συνάδελφο πρόεδρο της Επιτροπής ε, Τζούρι, τον κύριο Σβόμποντα, και να εκφράσω την χαρά μου που είμαστε σήμερα εδώ μαζί για αυτή τη σημαντική ακρόαση με εξαιρετικούς εμπειρογνώμονες. Συνεχίζω λοιπόν στα Ιταλικά. Πιστεύω πως είναι γνωστό πως η Επιτροπή Πολιτισμού από την προηγούμενη θητεία και συνεχίζοντας ε, παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τα θέματα και τις προκλήσεις ε, στα, στο, στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων όπου η δημιουργικότητα αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά τη νέα υπόθεση, όσον αφορά την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών, καθώς και την πρόκληση του, στην ψηφιακή, καθώς και το ίντερνετ. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ασχοληθεί πολύ με αυτό το θέμα, με γνώσεις και με γνωμοδοτήσεις που δώσαμε στο τομέα αυτό, όπως για την οδηγία για τα ορφανά έργα ή για την γενική προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και κυρίως για την online μουσική, αλλά σκέφτομαι και μία, ένα θέμα που αφορά αυτά εδώ τα προβλήματα, δηλαδή την ισορροπία που θα βασίζεται στην ιδιαιτερότητα του πολιτιστικού και οπτικοκουστικού περιεχομένου επιγραμμικά, καθώς και την διεύρυνση στην πρόσβαση στον πολιτισμό και στην πολιτιστική παραγωγή, την οπτικοστική από τη μια πλευρά και την ε, δίκαιη ανταμοιβή του ε, δημιουργού. Αυτά τα θέματα λοιπόν τα έχουμε συζητήσει πολύ στην Επιτροπή μας. Πιστεύω πως δεν μπορεί να υπάρχει ευρωπαϊκός χώρος πολιτισμού και δημιουργικότητας και στο πλαίσιο μιας της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και ισχυρός ανταγωνισμός ε, που μπορεί να προέλθει από την ανάπτυξη της ε, πολιτιστικής, ε, οπτικοακουστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, αν αυτά τα δικαιώματα δεν είναι εγγυημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό από αυτή την άποψη σημαντική μάλλον η εργασία που έχει γίνει όσον αφορά την προστασία, την προώθηση και την πρόσβαση στο on, στην online κληρονομιά, όπως αυτό το πρόγραμμα ε, το οποίο όλοι υποστηρίζουμε, το Ευρωπαίανα, καθώς και τη διασυνοριακή πρόσβαση στα επιγραμμικά περιεχόμενα. Άρα λοιπόν τα πνευματικά δικαιώματα σε μια ένωση όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται βασίζει μάλλον την ταυτότητά της στον πολιτισμό και στη δημιουργικότητα είναι εξαιρετικά σημαντικό ε, θέμα. Μετά από την ευρύτατη διαβούλευση στην οποία προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επί της οποίας είμαστε τώρα, ε, έχουμε τώρα μάλλον εγκύψει, Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να, έχουμε, να συμβάλλουμε για την σύσταση μιας νομοθεσίας που θα καλύψει αυτές τις ανησυχίες. Και είμαι ευτυχής που γνωρίζω πως έχετε επανεπιβεβαιώσει τη δημιουργία ομάδας εργασίας από την ομάδα Ζούρι που όπως στο παρελθόν ήταν πολύ κοντά ε, στους προγραμματισμού της Επιτροπής Πολιτισμού και είμαι σίγουρη ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί και να ευχαριστήσω και την κυρία Τρούπελ, η οποία ήταν εξέχον μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού την περασμένη θητεία και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο, έτσι ώστε αυτή η οδηγία να γίνει ε, μέσα από συνεργασία. Η σημερινή ακρόαση αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό στάδιο, γιατί έχουμε καλέσει ε, σπουδαίους ε, εμπειρογνώμονες για το θέμα αυτό και ευχαριστώ την γραμματεία της Επιτροπής Ζούρη και τον Προεδρό της που τους ε, καλέσατε και ελπίζω λοιπόν πως θα ολοκληρώσουμε αυτή την ε, αγαστή συνεργασία για το θέμα που αποτελεί πρόκληση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κώστα για τις παρατηρήσεις σας. Πρωτού δώσω το λόγο στον πρώτο μιλητή μας της ακρόασης να καταγράψω ότι ο Επίτροπος για την ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία, ο Γκίντερ Ρέτιγκερ, ανήγγειλε ότι μπορούμε να περιμένουμε από την πλευρά του την κατάθεση νομοθετικών προτάσεων σε ένα-δύο χρόνια. Αλλά ο Άντρου Σάντσιπ που είναι ο αντιπρόεδρος ο οποίος είναι αρμόδιος για την ενία αγορά είπε στην ακρόασή του ότι θα μπορούσαμε να αναμένουμε να δούμε προτάσεις στον τομέα αυτό μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Οπότε προσβλέπω σε μία διευκρίνηση από την κυρία Μάρτιν Πράτ, η οποία είναι και αρμόδια για τα θέματα τεχνολογίας, περιεχομένου, δικτύων πληροφορίας και copyright, θα μας δώσει μια καλύτερη διευκρίνηση για τα θέματα αυτά. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μου είπαν ότι πρέπει να κάθομαι κάπου εδώ. Δεν ήθελα να είμαι μακριά σας, όμως. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω επικροτώντας την πρωτοβουλία αυτή της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Πολιτισμού και Εκπαίδευσης για να έχουμε αυτή την πρώτη ακρόαση και ανταλλαγή απόψεων. Πρέπει να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινείται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι η Κομισιόν. Δεν θα ήταν σωστό όμως να πούμε ότι η Κομισιόν βραδιπορεί, γιατί η νέα Κομισιόν ασκεί τα καθήκοντά της μόνο για μια εβδομάδα και κάτι λίγο παραπάνω. Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων μου, τώρα εγώ δεν μπορώ να σας πω αν έχει δίκιο ο κύριο Σέτιγκερ ή ο κύριο Σάνσιπ. Αυτό είναι κάτι που αυτοί οι δύο μάλλον είναι σε καλύτερη θέση από μένα να σας απαντήσουν. Αλλά υπάρχει σαφής επίγνωση της ανάγκης να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα για τα θέματα αυτά. που αποτελούν και αυτά τα θέματα <clears throat> τμήματα των σαφών κατευθυντήριων γραμμών του Προεδρού Γιούγκερ. Αυτό το οποίο κάνουμε λοιπόν προς το παρόν είναι να βασιστούμε στο έργο το οποίο έχει επιτελεστεί τα τελευταία δύο χρόνια και όπως ξέρετε είναι μια σειρά από μελέτες νομικό-οικονομικού χαρακτήρα, ευρείες διαβουλεύσεις με τους εμπλεκομένους και υπάρχουν πολλές πολιτικές αποφάσεις που πρέπει εν καιρό να ληφθούν σε σχέση με το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης πρωτοβουλίας. Η Κομισιό φυσικά στη διάθεσή σας για να συζητήσει μαζί σας για τα θέματα αυτά μόλις ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει συνεργασόμενοι με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στο προηγούμενο Κοινοβούλιο ήταν πάρα πολύ καλή και με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή Πολιτισμού ήμασταν σε θέση να λειτουργήσουμε πάρα πολύ αποτελεσματικά για πολύπλοκα ζητήματα, πολλές φορές τεχνικού χαρακτήρα. Η κυρία Κώστα αναφέρθηκε στην ε, οδηγία για τα ορφανά εργατέχνης και επίσης και το θέμα των διαπραγματεύσεων για τη συνθήκη του Μαρακέσου. Είναι λοιπόν απόλυτα διατεθειμένη η Κομισιόν να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί σας όπως και την προηγούμενη θητεία για συζητήσεις τεχνικού χαρακτήρα και πολιτικού χαρακτήρα. Είμαστε στη διάθεσή σας λοιπόν. Με μεγάλη χαρά μπορούμε να είμαστε μαζί σας και να συζητούμε και τα πιο πολύπλοκα θέματα τα οποία μπορεί να θέλετε να συζητήσετε και είμαι σίγουρη ότι είσαστε έτοιμοι να συζητήσετε και τα αρμόδια πολιτικά θέματα με τον Επίτροπο και τον Αντιπρόεδρο που είναι υπεύθυνοι για τα θέματα αυτά στην Κομισιόν. Αυτά λοιπόν και εγώ έχω μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω αυτά τα οποία θα πούν οι εμπειρογνώμονες τους οποίους έχετε προσκαλέσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Ας περάσουμε τώρα στους προσκεκλημένους, προσκεκλημένους ειδικούς, εκ των οποίων Πρώτος είναι ο καθηγητής Μάρτιν Κρέτσμερ, καθηγητής του δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης. Έχετε το λόγο κύριε καθηγητά για 20 λεπτά. Καλησπέρα σας. Κύριε Συμπρόεδρε, Μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου και στην Νομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Πολιτισμού που οργανώνεται την ακρόαση αυτή που επιτρέπει έτσι μια ευρύτερη, προσέγγιση στη, στο νομοθετικό έργο. Έχω φτιάξει τώρα αυτή την ε, διαφάνεια που έχουν, ε, με τα όργανα που έχουν συνδημιουργήσει το κέντρο μας για πρώτη φορά μια εμπειρική προσπάθεια για τη μελέτη του δικαίου ε, βιομηχανικής ιδιοκτησίας από διάφορες πτυχές οικονομικές, κοινωνικές. Πρόκειται για ένα νέο είδος εγχείρημα που ελπίζουμε ότι θα προσφέρει κάποιες από τις που χρειάζονται οι νομοθέτες. Υπάρχουν συνολικά 40 ε, project, όλα αυτά εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ε, Επιτροπής σας. Ας αρχίσω σήμερα λοιπόν με μια σύντομη επανεξέταση των 20 χρόνων, 20 ετών κρίσης σε θέματα copyright. Βλέπετε τους τίτλους αυτούς που ε, ομαδοποιούνται ανανομικές παρεμβάσεις. Δεν είναι χρονολογική η σειρά δηλαδή. Κάποιες είναι σε διεθνές επίπεδο, κάποιες είναι σε εθνικό επίπεδο. Και βλέπει κανείς εδώ ότι ο προσανατολισμός έχει αλλάξει. Η πηξίδα έχει γυρίσει. Υπάρχει λοιπόν το ε, ψηφιακό θεματολόγιο με θέματα προστασίας, ξαναπάει να βάλει το τζίνι μέσα στο μπουκάλι και παρεμβάσεις που προωθούν περισσότερο την καινοτομία. Έχουμε διάφορες πρωτοβουλίες επιβολής και μετά άλλες πρωτοβουλίες οι προσπαθούν να επαναφέρουν κάποια ισορροπία. δεν θα εξετάσουμε σήμερα τα λεγόμενα cloud computing που είναι σημαντικά θέματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν και σε θέματα copyright αλλά θα εξετάσω περισσότερο στα 20 λεπτά που μου δίνετε την ε, μελλοντική, το μελλοντικό προσανατολισμό διότι μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί συνένεση. Θα μιλήσω ιδίως λοιπόν για τις τέσσερις ε, άβολες αλήθειες για το copyright που καμιά έρχονται σε σύγκρουση με πεπιθήσεις στις οποίες βασίζεται η πολιτική για το copyright οι οποίες πεπιθήσεις εμπειρικά αποδεικνύονται αμφίβολες αν όχι εσφαλμένες. Το πρώτο, η, η, πρώτη τέτοια πεποίθηση λέει ότι το copyright δεν εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια του καλλιτέχνου. Θα σας δώσω τις εμπειρικές ενδείξεις σε λίγο. Η δεύτερη τέτοια αρχή λέει ότι δεν μπορεί κανείς να αναγκάσει τον καταναλωτή να δαπανίσει χρήματα. Αντίθετο με την πεποίθηση που λέει ότι ο καταναλωτής είναι το πρόβλημα. Το τρίτο λέει non-use, μη χρήση πολλών έργων που εξακολουθούν να προστατεύονται από το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και αυτό πάλι έρχεται σε αντίθεση με την πεποίθηση ότι το copyright έχει την έννοια ότι θέλει να καταστήσει τα έργα αυτά πιο προσιτά στο κοινό και το τέταρτο λέει ότι η πολιτική copyright δεν έχει βάση βασισμένη σε ανεξάρτητες ενδείξεις. Σε δούμε λοιπόν την πρώτη από αυτές τις ε, άβολες αλήθειες. Ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια του καλλιτέχνη. Εμείς όλοι πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο είναι επενετό ως στόχος μιας πολιτικής. Σε πολλές παραθέσεις από νόμους που έχω βάλει εδώ, λέει ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η ανεξαρτησία και η αξιοπρέπεια του καλλιτέχνου και του δημιουργού είναι και μια πεποίθηση στην οποία βασίζεται η συνθήκη της Βέρνης η οποία αρχίζει απονέμοντας τα δικαιώματα στον δημιουργό και για τη διάρκεια της ζωής του. Αν δείτε όμως την εμπειρική πραγματικότητα των πολιτιστικών αγορών, η εικόνα που θα δείτε είναι μάλλον ενοχλητική. Έχουμε αγορές του είδους winner take all, ότι ο, αυτός που κερδίζει τελικά τα παίρνει όλα, δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, αλλά είναι γεγονός. Επίσης οι περισσότεροι δημιουργοί έχουν περισσότερες από μια πηγές εισοδήματος. Ε, τα global assignments, οι παγκόσμιες δηλαδή ε, διαθέσεις των δικαιωμάτων είναι κάτι το κοινό και φαίνεται ότι τελικώς η ιδιοκτησία των δικαιωμάτων δεν επιφέρει μεγάλη διαφορά. Με τις ε, διάφορε συμβάσει δηλαδή που υπογράφει ο δημιουργός αποχωρίζεται τα δικαιώματά του και αυτά μεταφέρονται σε άλλους. Αυτά μας βοηθούν να αντιληφθούμε τις ε, αγορές copyright ω αγορές εργασίας των καλλιτεχνών. Ως εσείς δηλαδή που ασκείτε την πολιτική θα έλεγα να είστε δυσπιστοί όταν έρχονται να σας μιλήσουν για τα δικαιώματα των δημιουργών. Να, να ρωτήσετε πρώτα να σας δείξουν τις συμβάσεις που υπογράφουν. Υπάρχουν βέβαια ανησυχίες για, τις, ε, για τα δικαιώματα των δημιουργών και για την προστασία των επενδύσεών τους. Αλλά να μην, να μην συγχαίονται τα συμφέροντα των εργαζόμενων και του κεφαλίου, όπως τα λέγαμε κάποτε. Αλλά εδώ χρειάζεται να γίνει διαχωρισμός των ενιών. Αυτό το winner take all ε, ως χαρακτηριστικό της αγοράς έχει και ένα δεύτερο στοιχείο. Είναι μια δομή όπου οι κληρονόμοι γίνονται δυσανάλογα σημαντικοί. Παράδειγμα, από την ε, οδηγία Resale Rights. όπου ο δημιουργός λαμβάνει ένα μέρος από το ποσό που ε, αποδίδει την υποπρασία και δείχνει η αλήθεια ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών καταλήγει στους κληρονόμους. Μόνο 18% καταλήγει στα χέρια δημιουργών που βρίσκονται ακόμα εν ζωή. Δεύτερο παράδειγμα, η παράταση των χρόνων διάρκειας. Πάλι βλέπουμε από το γεγονός και μόνο παράτασης του χρόνου μια μεταφορά από τους ζώντες δημιουργούς στους κληρονόμους. Γίνεται διαφορετική κατανομή της πίτας, δηλαδή έχουμε κάποια δεδομένα από τη Σουηδία που δείχνουν τι έγινε το 1995 όταν η Σουηδία προσεχώρησε και υιοθέτουν κανόνα το 50 συν Τα διάφορα κίνητρα πρέπει να αναφέρονται στους ζώντες ε, δημιουργούς. Αυτό το συναισθηματικό επιχείρημα του ε, καλλιτέχνη που πεθαίνει στην ψάθα πρέπει να το δει κανείς μέσα σε κάποια όρια το, το, τι, το τι πραγματικά σημαίνει δηλαδή στην αληθινή ζωή. Δεύτερο τώρα, θα πρέπει να σας ε, δώσω ίσως και κάποιες λύσεις. αντιμετωπίζοντας τις θεμητές ανησυχίες καλλιτεχνών και δημιουργών θα πρέπει να στοχεύσετε ιδίω σε συμβάσεις, σε ηθικά δικαιώματα και αποζημιώσεις που πρέπει να μπαίνουν και στις συμβάσεις και ίσως θα πρέπει να κατανοήσετε και τον τρόπο που λειτουργούν οι συλλογικέ εταιρείε εκπροσώπησης των δημιουργών. Ας έρθω τους καταναλωτές. Στη δεκαετία του 1990 προχωρήσαμε σε μελέτη για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας μουσικής και ήρθαμε σε επαφή με όλες τις μεγάλες εταιρείες τότε και η κυριαρχούσα στρατηγική τότε ήταν να περιφράσουν το περιεχόμενο σε ένα κλειστό κύκλωμα και να αναγκάζουν τον καταναλωτή να καταναλώνει μέσα σε αυτό το κλειστό κύκλωμα. Και το κύριο δικαίωμα ήταν το δικαίωμα να πει κανείς όχι. Ωστόσο, οι καταναλωτές αντέδρασαν. Άρχισαν να κατεβάζουν και να μεταφέρουν αρχεία και με καμία παρέμβαση δεν μπόρεσε να σταματήσει αυτό έως τώρα. Τα εμπειρικά στοιχεία που δείχνουν τώρα την στάση των καταναλωτών δείχνουν σαφώς ότι το κατέβασμα, downloading δηλαδή, και το share οδηγεί και σε περισσότερες πωλήσει. Αυτοί δηλαδή που κάνουν περισσότερο downloading καταναλώνουν και περισσότερο και αγοράζουν περισσότερα. Και το ζήτημα είναι πώς κατανέμεις αυτόν τον προπολογισμό ώστε να φτάσουν τα λεφτά από τον καταναλωτή στην τσέπη του δημιουργού. Αυτό πρέπει, να γίνει να κατανοήσουμε πώς δρούν οι καταναλωτές. Το να τους σφίξουμε ακόμη περισσότερο τα λουριά δεν πρόκειται να αλλάξει τη συμπεριφορά τους. Πρέπει να αντιληφθούμε πώς κάνουν τι επιλογές και υπάρχουν περισσότερα εμπειρικά στοιχεία που δείχνουν ότι αν το επιχειρηματικό μοντέλο μετατοπιστεί και οι υπηρεσίε προσφέρονται σε καλέ τιμέ στου καταναλωτέ, αυτοί αντιδρούν θετικά. Το δεύτερο εδώ για το ρόλο του καταναλωτή είναι ότι ο καταναλωτή θεωρεί το copyright σαν κάτι το οποίο καταναλώνει, αλλά μπορεί να είναι και εισρωή σε νέα έργα. Δεν θα ανοίξω εδώ όλη την σκηνή τώρα της δημιουργίας περιεχομένου, αλλά αυτό, σε αυτό καταλήγουν οι ερευνητές, δηλαδή ότι αυτό το input είναι και output, δηλαδή περνάει και στην έρευνα. Είναι σωστό να κατανοήσουμε το διαδίκτυο σαν κάτι παραπάνω από ένα μηχάνημα που βγάζει φωτοτυπίες ή που αντιγράφει απλά. Λύσεις. Έχει γίνει μεγάλη ε, πρόοδος ήδη προς την κατεύθυνση να, περάσει, να περάσουμε από τον καταναλωτή στην προσφορά των υπηρεσιών που να ενδιαφέρουν τον καταναλωτή. Και να εξετάσουμε και τις εξαιρέσεις από τις πρώτες αρχές. Δηλαδή ποιος είναι ο στόχος του δικαίου του copyright. Αν εξυπηρετεί ακόμη τους στόχους του. Εγώ πιστεύω ότι οι μη εμπορικέ χρήσεις είναι δυνατόν να υπάρξουν και θα πρέπει να τεθούν επιτάπητος. Η τρίτη άβολη αλήθεια είναι το copyright και η μη χρήση. Εδώ έχω στοιχεία από μια μελέτη του Paul Hild του Πανεπιστημίου του Ιλινόη τα πράγματα διαφορετικά από το 1950, από το 1950 μάλλον, και πρόκειται για ένα κλάδο ο οποίος κινείται ταχύτατα, έχει πολύ ταχύς κύκλους ε, προϊόντων, δεν μπορούμε να αναμένουμε δηλαδή ένα κενό και στο οποίο να επανέρχονται, γιατί τώρα επανήλθανε. Ε, έχουμε ένα κενό στο 1923, διότι οτιδήποτε πριν από αυτό είναι στο δημόσιο τομέα. Κάτι δεν λειτουργεί ωστόσο. Δεν υπάρχει υλικό διαθέσιμο που θα έπρεπε να υπάρχει. Εδώ υπάρχουν και άλλα δεδομένα για, τους, για τον κύκλο προϊόντων, δηλαδή υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα ένα ενδιαφέρουν. Τώρα λύσεις. όπως και με το δίκαιο των εμπορικών σημάτων, πρέπει να επιτευχθεί συνένεση πάνω σε μια πρώτη αρχή ότι τα δικαιώματα συνεπάγονται και υποχρώσεις. Δικαιώματα δηλαδή τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να συνεπάγονται κάποιες συνέπειες, ίσως όχι τόσο δρακόντιες όπως στον, στο δίκαιο περί εμπορικών σημάτων, που ένα εμπορικό σήμα εάν δεν χρησιμοποιηθεί για πέντε χρόνια τότε ανακαλείται, αλλά είναι πάντως δυνατό να αναπτύξει κανείς μηχανισμούς που θα επιτρέψουν την διάθεση έργου και μάλιστα σε αυτό να ωφελήσει και τον δημιουργό εφόσον επανέλθει το, το έργο σε αυτόν μετά από μια παραδοσμένου χρόνου χωρίς χρήση. Η τελευταία άβολη αλήθεια είναι πολιτική βασισμένη σε ενδείξεις evidence-based. Είχα ε, συμμετάσχει σε άλλη ακρόαση στην Επιτροπή σας για ηχογραφήσεις και τις σχετικές ε, διατάξεις προστασίας των δικαιωμάτων και έχω και ένα άθρο από εκείνη την οδηγία. Ήταν μια ρήτρα η οποία φάνηκε αθώα τότε. Με τα λόγια που λέει shall expire, θα εκπνέουν δηλαδή 70 χρόνια μετά τον θάνατο του τελευταίου προσώπου κλπ. Ο συγγραφέας των στίχων δηλαδή και ο συνθέτης της μουσικής εφόσον η συνεισφορά τους ήταν ειδική για το συγκεκριμένο έργο. Αυτό φαίνεται να είναι μια απλή εναρμονιστική διάταξη, αλλά από τότε έχει καταστεί σαφές ότι πίσω από αυτό κρυβόταν κάποιο λόμπι. Και μπορώ να σας δείξω και το παράδειγμα. Ο George Γκέρσον πέθανε το 1937, ο αδελφός του πέθανε το 1983 και με αυτή τη μικρή ρήτρα που λέει ο τελευταίος νομοθέτης, ο προηγούμενος νομοθέτης, δηλαδή το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψαν ώστε η κληρονομιά των Γκέρσουιν να δημοπρατηθεί και επομένως ευρωπαϊκά χρήματα να καταλύσουν σε non-practicing entities. Ίσως ως νομοθέτες να μην να θέλουμε να εξετάσουμε σε βάθος τα τις πριν να λάβουμε απόφαση. τέλος, κάτι που έχει συζητηθεί σε πολλά βήματα, η διαπραγματευτική θέση της Ένωσης στην ΒΑΙΠΟ και στη βάση της οποίας διαφορετική πολιτική ακολουθείται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι σε διεθνή φόρα και όπου πάλι εδώ πιστεύω ότι μια ορθή πολιτική βασισμένη σε ενδείξεις πρέπει να γίνει με τρόπο διαφανή. Συμπέρασμα τώρα. για την ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια του καλλιτέχνη. Προστασία δικαιωμάτων, δημιουργών κλπ. Δυστυχώ ο διαφάση διαβάζει κείμενα με ταχύτητα και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Είτε πρόκειται για θα πρέπει να υπάρχει με εμπειρικό τρόπο καθοδήγηση του πλαισίου. Για τη μη χρησιμοποίηση υπάρχει πολύ υλικό το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το οποίο αλλιώς θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν οι καινοτόμοι καλλιτέχνες. Τέταρτον, μια πολιτική η οποία να βασίζεται σε στοιχεία. Σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλά από αυτά τα θέματα βελτιώνεται η γνώμη μας, η γνώση μας. Έχουμε πολλές ανεξάρτητες μελέτες οι οποίες μπορεί να μας βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτή τη στιγμή το copyright βοηθάει αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλες συλλογέ από ε, κληροδοτήματα με αρνητικές συνέπειες. Αυτό θα πρέπει να ανατραπεί με το να μπορέσουμε να προωθήσουμε μια πιο ζωντανή δημιουργική Ευρώπη. Το παράδειγμα Γκέρσουιν δείχνει ότι κάθε παρέμβαση εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα περισσότερο από άλλα. Αν η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει ένα ηγετικό ρόλο στην πολιτική copyright, θα πρέπει να κάνει σημαντικές αλλαγές. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία για την ανάγκη να ασκήσουμε πολιτική. Ευχαριστώ σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Τα επόμενα 20 λεπτά θα τα αναλάβει ο καθηγητής Τόμπους, ο οποίος είναι καθηγητής ε, στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Έχετε το λόγο κύριε καθηγητά. Σφόμποντα, κυρία Κώστα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε για να σας ε, παρουσιάσω κάποιες σκέψεις και μια σύντομη μελέτη που έκανα για την έκθεση αυτή που αφορούσε τον, ε, τη διαβούλευση της τελευταίας Επιτροπής για τα θέματα copyright. Ξεκινώ με το να εκφράσω την ε, εκτίμησή μου για αυτά που είπε ο κύριος Κρέτσμερ προηγουμένως, ο προλαλής σας. Δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο μαζί του, τόσο σε ό,τι αφορά την ουσία, αλλά και σε ό,τι αφορά το επίκαιρο αυτής της ακρόασης, στη δική μου περίπτωση. Πιστεύω ότι ενώ υπάρχει μια νέα επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντα της λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν, ίσως είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία έχει επιτύχει η προηγούμενη Κομισιόν σε σχέση με τη δημόσια διαβούλευση για το copyright και την έκθεση που εξέδωσε αυτή η Επιτροπή. Ακριβώς σε αυτό θα εστιάσω τώρα στην ομιλία μου. Ξεκινώ με το να εξηγήσω γιατί ασχολούμαι με την έκθεση της Κομισιόν. Καταρχήν, παρά το γεγονός ότι το δίκαιο του copyright είναι και φυσικά το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο νομικό ζήτημα, υπάρχει μια βασική γραμμή με την οποία όλοι μπορούν να συμφωνήσουν. Ότι το copyright είναι μια επιζήτηση ισορροπίας. Και αυτός είναι και ο τίτλος ενός εισαγωγικού εγχειριδίου για το copyright. Το πρώτο του κεφάλαιο έχει αυτόν τον τίτλο και έχει γραφτεί από τον Άλαν Κιλ Πάτρικ. Θα έλεγα επίσης ότι είναι διπλά ε, επιζήτηση εξισορρόψης, διπλή ισορροπία. Από τη μία πλευρά θα πρέπει να εξισορροπήσει την πρόσβαση και την προστασία. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε προηγούμενα έργα, δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία έκφρασης και θα μαραθεί η δημιουργικότητα. Χωρίς προστασία όμως πολλά μοντέλα επιχειρηματικά βασίζονται στο copyright θα καταστρεφόντουσαν. Γι' αυτό το λόγο ο Μάρτιν Κρέτσμερ προηγουμένως σας παρουσίασε την ε, προβληματική αυτή. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με αυτά τα ουσιαστικά θέματα. Θα ασχοληθώ περισσότερο με το δεύτερο πρόβλημα ισορροπίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους νομοθέτες γιατί πρέπει να εξορροπήσουμε τα συμφέροντα των εμπλεκομένων, τα οποία πρέπει να εξορροπήσετε ως νομοθέτες. Έχω τονίσει ιδιαίτερα την ε, ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των εμπλεκομένων και αυτό βασίζεται και στις, στην ε, έκθεση της Κομισιόν για τις απαντήσεις στη δημόσια διαβούλευση για τη μεταρρύθμιση των κανόνων του copyright στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση κάνει εύκολη την ανάλυση γιατί ζητήθηκε στην διαβούλευση οι απαντώντες να πούν σε ποια κατηγορία εμπλεκομένων βρίσκονται. Κυρίως ήταν καταναλωτές, ήταν οι δημιουργοί, οι ερμηνευτές, ήταν πάροχοι υπηρεσιών, ήταν συλλογικοί οργανισμοί διαχείρισης κτλ. Βέβαια, ο αριθμό των απαντήσεων ήταν άνισα κατανοημένο μεταξύ των ομάδων αυτών των εμπλεκομένων Πήραμε περίπου 11.000 απαντήσεις, οι περισσότερες όμως προέρχονται από τους ε, ε, δημιουργούς, αλλά επειδή η έκθεση έχει να κάνει με τις απαντήσεις των ε, ε, εμπλεκομένων, δεν υπάρχει έλεγχος του αριθμού των απαντήσεων, απλώς προσπαθεί η Κομισιόν να καταλήξει σε, μια συλλογική εικόνα. Λόγω αυτής της πολλαπλότητος των εμπλεκομένων, τι θα πει εξισορρόπηση για το copyright. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε σαφές ο Μάρτιν Κρέτσμαν. Δεν είναι μονάχα η βιομηχανία εναντίον των καταναλωτών. Υπάρχουν διάφορα εμπλεκόμενοι, διάφορα συμφέροντα σε διαφορετικές καταστάσεις. Θα έλεγα ότι η εξισορρόπηση στα θέματα του copyright σημαίνει εξέβρεση μιας συμβαστικής λύσης και θα μπορούσαμε να έχουμε μια ευριστική διαδικασία η οποία κάνει τη συνένεση στην περίπτωση που όλοι είναι εξίσου δυσαρεστημένοι. Δεν είναι επιστημονική αυτή η προσέγγιση, είναι μια δοκιμαστική αντιμετώπιση, αλλά αυτό θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε δύο ερωτήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το νόμο του copyright. Το πρώτο ερώτημα είναι πόσο εξισορροπημένη ή μη εξισορροπημένη είναι η τωρική, τωρινή νομοθεσία για το copyright στην Ευρώπη. Λέω ο Μάρτιν Κρέτσμε ότι δεν υπάρχει ισορροπία εκεί. Αλλά τι λέει η έκθεση διαβούλευση για τα θέματα αυτά και πώς την αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι. Παρά το γεγονό ότι το ευρωπαϊκό copyright δεν έχει αλλάξει μετά από την έγκριση αυτή τη οδηγία, η ισορροπία μπορεί να έχει αλλοιωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία λόγω των τεχνολογικών αλλαγών, παραδείγματο χάρη. Αυτό δεν είναι τίποτα το παράξενο όταν περάσαμε από την μουσική, την καταγεγραμμένη ε, σε δίσκους η οποία πολλές φορές απίτησε μια όταν περάσαμε στο ίντερνετ υπήρξε μια σημαντική αλλαγή τεχνολογίας η οποία πολλές φορές απίτησε μια επανεξισορρόπηση νομοθεσίας. Δεύτερον, εάν δούμε ότι δεν υπάρχει επαρκής ισορροπία στο δίκαιο του copyright, τι πρέπει να κάνουμε για να επαναφέρουμε αυτή την ισορροπία προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν οι προσπάθειες επαν εξής ορόπησης. Για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, έχω επανεξετάσει την πρόταση της Κομισιόν για τη δημόσια διαβούλευση. 100 σελίδες σύνοψης, 9.500 απαντήσεων και 11.000 υπεραιτέρω μηνυμάτων. Μια έκθεση η οποία ακολουθεί τη δομή του ερωτηματολογίου που τέθηκε στο διαδίκτυο με 80 ερωτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε 24 τμήματα. Για κάθε μία από αυτές τις ε, πτυχές ε, η έκθεση διακρίνει την απάντηση 9 ομάδων εμπλεκομένων. Εγώ στην έρευνά μου κοιτάω για κάθε μία ένα από τα 24 θέματα αν οι έξι κέρυες ομάδες των ε, εμπλεκομένων που είναι οι τελικοί χρήστες και καταναλωτές, θεσμικοί χρήστες, η παροχή υπηρεσιών και η ενδιάμεση, η δημιουργοί και οι ερμηνευτές, οι οργανώσεις συλλογικής διαχείρισης και οι εκδότες ε, και εκπομπή, κανάλια κτλ. Αν ήταν ικανοποιημένοι ή όχι με το περιεχόμενο της νομοθεσίας. Έχω χρησιμοποιήσει χρώματα, πράσινο χρώμα για ικανοποίηση, μάλλον πράσινο χρώμα αν θέλουν κάποια μεταρρύθμιση, αν υπάρχει κάποια τέτοια ε, πρόταση που κάνουν για αλλαγή. Κόκκινο σημαίνει ότι δεν θέλουν καμία αλλαγή, είναι ικανοποιημένοι με το status και δεν βλέπουν καμία ανάγκη αλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κίτρινο, στην περίπτωση που δεν είναι σίγουροι οι, αυτοί που απαντούν ή θεωρούν ότι το θέμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με το copyright. Συγκεκριμένο παράδειγμα, ένα θέμα παραγωγής χάρη το οποίο αντιμετωπίστηκε από δύο ερωτήματα ήταν η εδαφικότητα των εξαιρέσεων για το copyright. Εδώ βλέπετε ότι οι τελικοί χρήστε και οι θεσμικοί χρήστες, βιβλιοθήκες, μουσεία κτλ. βλέπουν προβλήματα και την ανάγκη να υπάρξει μια σειρά από κανόνες ενώ οι ενδιάμεσοι έχουν μια διαφορετική άποψη εδώ και κάποιοι άλλοι, οι ερμηνευτές και οι δημιουργοί θεωρούν ότι δεν είναι πρόβλημα η ιεραρχικότητα. Ένα άλλο παράδειγμα, αν κοιτάξτε το θέμα των νέων εξαιρέσεων, παραδείγματος χάρη το θέμα της εξόριξης κειμένου και δεδομένων. Υπήρχε εδώ η ανάγκη να υπάρξει κάποια, κάποια μορφή περιορισμού στην οδηγία αυτή οι τελικοί χρήστες καταναλωτές και οι θεσμικοί θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να γίνει μια τέτοια αλλαγή, ενώ οι οργανώσεις συλλογικής διαχείρισης, οι ερμηνευτές και οι ε, δημιουργοί δεν το θεωρούν ότι είναι έτσι τα πράγματα. Σε ορισμένε περιπτώσει όμως δεν υπάρχει αυτή η ε, οριοθέτηση μεταξύ των απόψεων. Παραγωγή χάρη στο θέμα της ε, δίκαιας αμοιβή των ερμηνευτών και δημιουργών οι ομάδες αυτές και οι δημιουργικοί οι ερμηνευτές αλλά και οι καταναλωτές θεωρούν ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει νομοθετική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η δίκαια ανταμοιβή των καλλιτεχνικών δημιουργών. Και αυτό ε, πιστεύω ότι έχει να κάνει και με αυτά τα οποία ανέφερε ο Μάρτιν Κρέσμε που έχουν να κάνουν με τη συλλογική διαπραγμάτευση για τα συμβόλια. Ενώ οι ενδιάμεσοι και οι εκδότες δεν βλέπουν ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτά είναι συγκεκριμένα παραδείγματα τώρα. Αν δούμε τώρα την συνολική εικόνα, τη μεγάλη εικόνα που προκύπτει από αυτή την ανάλυση και δείτε και τα 24 τέτοια θέματα και το κατά πόσο οι ομάδες των εμπλεκομένων ήταν υπέρ ή κατά της μεταρρύθμισης. Βλέπετε αυτή την εικόνα, δεν είναι κάπως, δεν είχε πολύ εκπληκτικό το αποτέλεσμα. Είναι σαφές ότι έχουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ των ε, εμπλεκομένων. Οι τελικοί χρήστες και οι θεσμικοί χρήστες είναι από τη μία πλευρά και υποστηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις, ενώ η παραγωγή, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι δημιουργοί και ερμηνευτές προτιμούν το τωρινό σύστημα όπως είναι. σε 22 ή 23 περιπτώσεις θέλουν τελικοί χρήστες και θεσμικοί χρήστες αλλαγή, ενώ από την άλλη πλευρά η παραγωγή και οι διαχειριστές συλλογικών συλλογών θεωρούν ότι πρέπει να παραμείνει στις right ως έχει αυτή τη στιγμή. Επίσης, διστακτική για τη μεταρρύθμιση είναι οι, οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές. Έρχομαι λοιπόν στα δύο αρχικά μου ερωτήματα. Δείχνει αυτή η ανάλυση ότι το ευρωπαϊκό σύστημα copyright είναι μονόπαντο. Δεν είναι εξισορροπημένο. Όταν μια πλευρά είναι ικανοποιημένη με το status quo και η άλλη είναι πολύ δυσαρεστημένη, αυτή δεν είναι μια εξισορροπημένη κατάσταση. Προς τα πού θα πρέπει να κινηθεί λοιπόν η προσπάθεια επανεξισορρόπησης. Νομίζω ότι από αυτή τη ε, μελέτη μπορούμε να μάθουμε κάτι για την κατεύθυνση επανεξισορρόπησης και αυτό δεν είναι μια βολική αλήθεια γιατί πρέπει να πάρουν μια συγκεκριμένη θέση οι νομοθέτες. Η επανεξισορρόπηση δεν πρόκειται να ικανοποιήσει όλο τον κόσμο, θα πρέπει να κάνει όλο τον κόσμο εξίσου δυσαρεστημένο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση κάποιας μεταρρύθμισης όπως ζητούν οι τελικοί χρήστες και οι θεσμικοί χρήστες. Και αν θέλετε να μπείτε στις λεπτομέρειες, τα στοιχεία βρίσκονται στην διεύθυνση αυτή. Δεν χρειάστηκα τα 20 λεπτά μου, αλλά νομίζω ότι έχετε καταλάβει τι ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Uh, we thank you, uh, και εμείς ευχαριστούμε κύριε καθηγητά για τα ενδιαφέροντα δεδομένα και στοιχεία που θέσατε υπόψη μας και να δώσουμε το λόγο τώρα για άλλα 20 λεπτά στον κύριο Μπουράκ Οσγκέν σύμβουλο της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εταιριών Δημιουργών και Συνθετών. Μάλιστα, ευχαριστώ τις δύο επιτροπές σας που οργανώσατε την ακρόαση και που μας προσκαλέσατε. Φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις διαφάνειες. Να σας εξηγήσω πρώτα ποιοι είμαστε. 34 γραφεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάνω από ένα εκατομμύριο ε, δημιουργούς και κατόχους δικαιωμάτων και στη μουσική και σε άλλους κλάδους δημιουργίας. Και οι εταιρείε μας ανέρχονται στο 36%, στο 61% μάλλον των εσόδων. Θα δείτε εγώ ήθελα μάλλον να αρχίσω την παρέμβασή μου με τις απόψεις των ίδιων των δημιουργών για το δίκαιο της ε, ιδιοκτησίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Και τους ρωτώ κιόλας ε, τι σημασία έπαιξε το copyright στην καριέρα τους. Θα ακολουθήσει από ό,τι αντιλαμβάνεται για μέσα ένα μικρό βίντεο το οποίο δεν πρόκειται να μεταφραστεί. No. Then I was hired to do a song for Eurovision and we won the Finnish entry and so forth. And then I started thinking that, you know, maybe I could live by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 Εμείς θέλαμε να ακουστεί πραγματικά η φωνή των καλλιτεχνών. Αλλά δυστυχώ για τεχνικού λόγου δεν έγινε δυνατό αυτό. Αρχικά όμω όταν το είχαμε δοκιμάσει λειτουργήσε το σύστημα. Τώρα δεν λειτουργήσε. Μήπω μπορούμε να επανέλθουμε τώρα στην ίδια την παρουσίαση. Τι να κάνουμε λοιπόν. στο φιλμ βλέπει κανείς πολλούς καλλιτέχνες που λένε το copyright πόσο σημαντικό ήταν για τη ζωή τους και για την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Και αυτό μιλεί από μόνο του. Αντί να περνάμε μέσα από κάποιες μελέτες και ξανά έρευνες και μελέτες που είναι και λίγο πολύ εξυπηρετούν ένα αυτοσκοπό να αποδείξουν κάτι από την αρχή δηλαδή. Ενώ το copyright είναι απαραίτητο για να συνεχίσει να δημιουργεί ο τομέας. Και ο κλάδος copyright είναι και μεγάλη πηγή εισοδήματος για όλο τον κλάδο. 56% των Ευρωπαίων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πολιτιστικούς σκοπούς. 9 από 10 παρακολουθούν βίντεο που έχουν σχέση με μουσική στο YouTube και 90% παρακολουθούν βίντεο από το διαδίκτυο. Είναι τεράστια πηγή ε, για, τα πλονεκτήματα προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Πρέπει να εξετάσουμε τον εκθετικό παράγοντα με τον οποίο ε, προχωρεί ο πολιτισμός και αποδίδει στην ψηφιακή οικονομία. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Χρειαζόμαστε ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα του δημιουργού, για το copyright. Είναι προτεραιότητα για να επιβιώσει η ο κλάδος της ψηφιακής οικονομίας. Ακούμε συχνά ότι οι καταναλωτές θέλουν πρόσβαση στο δημιουργικό έργο από παντού και οποτεδήποτε. Αυτό είναι σημαντικό νέο. Αυτό χρειάζεται πολυεδαφική άδεια, ε, διαθεσιμότητα διασυνοριακή και δυνατότητα μεταφοράς, portability δηλαδή. Βλέπουμε αυτό το multi-territorial licensing. Μόλις τώρα εγκρίναμε ε, οδηγία για την διαχείριση με, που περιλαμβάνει και το multi-territorial για τα μουσικά έργα και άδειες και άδειες δηλαδή διασυνοριακές και, εδαφι, και πολυεδαφικές. Αυτά προς όφελος όλων. Είδαμε επίσης στην πρωτοβουλία του 2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής License for Europe το Music Subgroup που σταμάτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι δεν υπήρχαν επαρκές, επαρκείς λύσεις στην αγορά και χρειάστηκε να συνεχιστούν οι συζητήσεις για το θέμα αυτό. Υπάρχουν 300 επιγραμμικές υπηρεσίες ε, μουσικής με πολλά ε, εκατομμύρια ε, τραγουδιών και κομματιών που προσφέρονται. Και το online arts είναι μακρά επιτυχία. Και έχουν τη διάθεση οι operator να επενδύσουν εφόσον δοθούν οι σχετικές άδειες. Και σύμφωνα με την έκθεση της, του Ευρωπαϊκού Ακουστικού Παρατηρητηρίου υπάρχουν 3.000 υπηρεσίες video on demand στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δούμε τώρα και τη διαθεσιμότητα διασυνοριακά, από εμά αυτό που κάνουμε τώρα είναι κοιτούμε τον αριθμό πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, τις υπηρεσίες βασισμένες στο νέφος, πρόσφατα έχουμε υποβάλει συστάσεις με δημόσιους σταθμούς για να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους και διαμεθοριακά και είμαστε και σε επαφή και με το εμπορικό ραδιόφωνο για να πετύχουμε παρόμοια συμφωνία. Βλέπουμε επίσης, μας δείχνει δηλαδή η πραγματικότητα της αγοράς ότι είναι περιορισμένη η αγορά ή αλλάζει ανάλογα με το περιεχόμενο. Τα πιο δημοφιλή ρεπερτουάρ μας είναι γαλλικά, γερμανικά και βρετανικά. Γαλλικό, γερμανικό και βρετανικό δηλαδή. Που έχουν 30 διαμεθοριακές ε, ε, άδειε ενώ το σλοβακικό μηδέν και ούτω καθεξής. Όλη η ανάπτυξη πανευρωπαϊκά έχουν ήδη κατακτήσει την αγορά και εγώ προτιμώ να στοχεύσω στα διάφορα ακροατήρια για να μπορέσω να αυξηθώ και συλλογικές άδειες είναι η σωστή συνταγή για να επιτύχουμε να προσεγγίσουμε τα ακροατήρια αυτά. Και ό,τι αφορά τώρα το portability, μπορεί κανείς να περάσει από φορείς όπως Spotify, Deezer, iTunes κτλ και να δημιουργήσει λογαριασμούς εκεί. Περνούν οι υπηρεσίε αυτές από εμά πρώτα και μετά αποφασίζουν πώ θα διανύμουν τα έργα του. Το ίδιο ισχύει και για τι εικαστικέ τέχνες, για ηλεκτρονικά βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες κτλ. Και είδαμε πάλι στο Licenses for Europe, στον οπτικό-ακουστικό τομέα, κοινή δήλωση για διασυνοριακές υπηρεσίες. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι χρειάζεται να βασιστούμε πάνω σε αυτές τις συνεχιζόμενες εξελίξεις αντί να αρχίζουμε ξανά από την αρχή κάθε φορά. Και ιδίω όταν βλέπουμε καθαρά τους λόγους που έχουν επίπτωση στην πανευρωπαϊκή παροχή υπηρεσιών, υπηρεσιών που βασίζονται σε επιλογές, επιχειρηματικές επιλογές. Το Spotify στην Ιταλία άρχισε πριν από δύο χρόνια όταν πέρασε από όλες τις ε, απαραίτητε άδειες. Δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο όσο στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βλέπουμε επίσης το roaming ή την, ε, τις διασυνδέσεις ε, ευρέως φάσματος και επίσης τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές πληρωμές. Και κάτι που βλέπουμε όλο και περισσότερο είναι εργατικό δίκαιο και προβλήματα φορολογικά που αποτελούν πολύ σημαντικό κόλλημα για ε, διάφορες επιχειρήσεις που αρχίζουν να λειτουργούν τώρα, startups δηλαδή. Άλλη δήλωση, statement B, είναι ότι οι άνθρωποι θέλουν ε, ε, ευκολότερη πρόσβαση σε διάφορα πολιτιστικά και άλλα έργα που επιθυμούν. Η αγορά δημιουργείται με δύο τρόπους. Αφενός με επιχειρήσεις, startup και υπηρεσίες που έχουν ακρόαση on demand κλπ όπου υπάρχει σχετική αδειοδότηση στην αγορά. Από την άλλη μεριά υπάρχουν άτομα ή χρήστες μικρής κλίμακας όπου πάλι υπάρχουν διαθέσιμα συστήματα μικρών, μικρά συστήματα χορήγησης αδειών που υπάρχουν community projects ή μικρές επιχειρήσεις η ε, χρήση ε, μουσικής ως background κλπ. Και υπάρχουν βεβαίως και όλοι οι θεσμικοί χρήστες είτε πρόκειται για σχολεία, είτε πρόκειται για πολιτιστικούς οργανισμούς κλπ. Και εκεί έχουμε εμείς να προσφέρουμε κάποιες επιλογές και έχουμε και, τα, και τους ήχους Ευρωπαϊκά που τους προσφέρουμε στο διαδίκτυο με τη συμμετοχή της Βρετανικής Βιβλιοθήκης και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς. Με λίγα λόγια προσπαθώ να πω ότι δεν χρειάζεται να αποδυναμώσετε τα δικαιώματα των δημιουργών για να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας. Αυτό που χρειάζεται είναι απλή συμπεριληπτική πρόσβαση, συλλογικές άδειες και μέσω συνεργασίας να γίνουν οι κανόνες πιο εύκαμπτοι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα περισσότερα από τα θέματα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τώρα και σε σχέση με τις ε, εταιρείες κλπ ακούμε την φράση τώρα επικοδομητική καταστροφή ή δημιουργική καταστροφή ως λόγο για να υπάρξουν νέα μοντέλα που θα αποδυναμώσουν το copyright. Αλλά να ξεκινήσετε ένα οικονομικό μοντέλο από μια καταστροφή δεν είναι σωστό. Δηλαδή καταστρέφεται αυτούς που προσφέρουν στην αγορά. Ενώ χρειάζεται αλλαγή του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζεται το κοινό μια εγγύηση που θα λέει μονάχα take and deliver χωρίς να εξασφαλίζουν την ε, συνένεση του δημιουργού θα καταλήξει σε τελικά σε καταστροφή της ίδιας της βάσης προσφοράς στην αγορά. Ενώ είναι νόμιμες επιχειρήσεις αυτές οι οποίες πληρώνουν τους φόρους τους και λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του νόμου. Γι' αυτό η συνένεση και η ανταμοιβή δεν έγινε το λεγόμενο ε, αποτέλεσμα παγώματος, το chilling effect χρειάζεται χρήση της τεχνολογίας με αποζημίωση των δημιουργών έτσι ώστε να υπάρχει βιώσιμη επιλογή σε κόστος που να μπορεί να το αντιμετωπίσει ο καταναλώτης. Σημαντικό, σημαντική επίσης είναι η συλλογική διαχείριση διότι διευκολύνει την χορήγηση συνένεση με νομική ασφάλεια αντιμετωπίζοντα τι πραγματικές ανάγκες των δημιουργών και καλλιτεχνών. Ποιε είναι οι άλλες τώρα προκλήσεις για μια ε, ισορροπημένη ψηφιακή οικονομία. Υπάρχουν θέματα τα οποία μας απασχολούν και πάλι εμείς θέλουμε προστασία των δημιουργών και ε, ε, θα τους ακούσουμε τώρα και ελπίζω πράγματι να μπορούσαμε να τους ακούσουμε στο φιλμ. That, um, I think we... Είναι τόσο σημαντική. Uh, as creators, as authors, we need to be very proactive in engaging in seeing where the value in that system is because um,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 δεν μπορούμε τελικά να ακούσουμε τη φωνή των δημιουργών. Δύο πράγματα ζητούμε και θα τα πω πολύ σύντομα. Πρώτον, διατήρηση και προώθηση της ορθής αξιοπρεπούς αποζημίωσης των δημιουργών και κυρίως από νέες πηγές για το private coping. Το κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση για την αντιγραφή που διατηρεί τον κύκλο αυτό. Το άλλο είναι όταν μιλούμε για copyright είναι κάπως σαν τον ελέφαντα μέσα στην αίθουσα που δεν τον βλέπει κανείς και ακούσαμε πριν ορισμένους δημιουργούς που λένε ότι πρέπει να αντισταθμίσει η από να η απώλεια αξία στη ψηφιακή οικονομία που σημαίνει ότι υπάρχουν online intermediaries οι οποίοι εποφελούνται αποκομίζουν τεράστια ωφέλη από τα δίκτυα και τις πλατφόρμες τους χωρίς να αναλαμβάνουν ωστόσο απολύτως καμιά ευθύνη για θέματα copyright και για αμοιβέ. Κρύβονται πίσω από το καθεστώς της e-commerce directive. Και γι' αυτό θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί πρέπει να ηγηθούν της συζήτηση. Το ίδιο είπαμε και στην δήλωση που υπέγραψαν οι δημιουργοί μας για μια Ευρώπη που θα δημιουργήσει απασχόληση. Αν έχετε ρωτήσει εδώ είμαι. Σας ευχαριστούμε για τις απόψεις σας. Μήπως μπορείτε να κλείσετε το μικρόφωνο σας. Τώρα το λόγο θα πάρει η κυρία Ιζαμπέλ Φέλτμαν, που είναι αναπληρώτρια γενική γραμματέας του οπτικοακουστικής λέσχης του Παρισιού. Είναι εμπειρογνώμονα ε, για θέματα πνευματικής διοκτησία, στους τομείς των τεχνών και της λογοτεχνίας, των οπτικοακουστικών και του ενοχικού δικαίου. Καλημέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Νομική Επιτροπή και την Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού που με κάλεσαν για να εκφράσω τη γνώμη μου ε, για αυτή την ανάλυση πολύ σημαντική εν ώψη της ενδεχόμενης αναθεώρησης των πραγματικών δικαιωμάτων μετά από αυτήν τη δημόσια διαβούλευση. Πριν να κάνω την παρέμβασή μου, μετά από τα όσα ακούσαμε, έχω την εξή παρατήρηση να κάνω. τα πνευματικά δικαιώματα είναι ένα δικαίωμα ιδιοκτησία, ιδιοκτησιακό δικαίωμα και είναι πολύ θεμελιώδε. Υπάρχει μια έλλειψη ισορροπία γιατί αυτό που δεν είναι σωστό είναι ότι τα συμφέροντα του δημιουργού και τα συμφέροντα του επενδυτή είναι ανακατεμένα. Είναι πολύ καλό να είναι έτσι ανακατεμένα τα συμφέροντα του δημιουργού και του επενδυτή από τη μια πλευρά. Γιατί όταν εργάζεται κανεί σε αυτό το τομέα, στη μουσική ή στα οπτικοακουστικά, ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα δημιουργό από μόνο του δεν μπορεί να δώσει μορφή στη δημιουργία του χωρί έναν επενδυτή ή του επενδυτέ. Δηλαδή, ποιοι είναι, είναι η παραγωγή, είναι οι διανομή, οι διαφημιστές και διαφορετικά ε, η δημιουργία αυτή θα έμενε κάτι ε, το ιδεατό που δεν θα μπορούσε να είναι προσβάσιμο για τους καταναλωτές. Ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει, λοιπόν, να θεωρείται λοιπόν ε, έλλειψη ισορροπίας. Είναι μάλιστα αντίθετα αυτό ε, ένα είδος αλληλεγγύης που δημιουργείται μέσω αυτής της αλυσίδας και από αυτήν εξαρτάται η επιτυχία μιας δημιουργίας και η πρόσβαση σε αυτήν ενός μεγάλου αριθμού καταναλωτών. Αυτά σε σχέση με τόσα είπαν οι προηγούμενοι ε, ομιλητές Φλέτσερ και Ντεμπούρ. Η δημόσια διαβούλευση και η έκθεση αυτή έχουν ε, προκαλέσει πολλά θέματα και διακυβεύματα όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Τρία συγκράτησαν την προσοχή μου και καταρχήν. Καταρχήν το πνευματικό δικαίωμα, πώς αυτό ε, ε, θεμελιώνεται σε μια κινούμενη και εξελισσόμενη αγορά. Ε, δεύτερον, η εδαφικότητα των δικαιωμάτων είναι δυσκολία για την πρόσβαση ή όχι. Ε, οι καταναλωτέ δηλαδή έχουν δίκιο να λένε ότι πρέπει να μεταρρυθμιστούν τα πνευματικά δικαιώματα λόγω τη εδαφικότητα των δικαιωμάτων αυτών. Και έπειτα, τρίτον, Ποια λύση θα μπορούσαμε να βρούμε για να ανταποκριθούμε σε αυτό το έντονο και σημαντικό αίτημα των δημιουργών και στη σχέση αυτή που έχουν μέσα στο πλαίσιο ε, τη σύμβασή τους με τον παραγωγό, αλλά που λόγω της εκμετάλλευσης αυτών των έργων τους σε μια ψηφιακή αγορά που έχει τεράστιο, ε, τεράστια εμβέλεια και μέγεθος. Το δικαίωμα, η εδαφικότητα λοιπόν και οι ενδεχόμενες επιπλέον αμοιβέ το πνευματικά δικαιώματα στην Ευρώπη είναι εναρμονισμένα μετά από την ανακοίνωση της 19 η Μαΐου 2010, στρατηγική, ψηφιακή στρατηγική στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες αλλά και προέβησε σε νομοθετικά μέτρα γιατί το είδαμε και πριν από λίγο ότι έχουν εκδοθεί διάφορες οδηγίες, ε, οδηγία για τη διάρκεια των δικαιωμάτων, για τα ορφανά έργα, για την ε, ε, συλλογική διαχείριση. Πρόκειται δηλαδή για ένα κοινό, μια κοινή βάση ε, για τις εθνικές νομοθεσίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ε, πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Είναι λοιπόν πολύ στέρεη αυτή η νομοθεσία συμπαγής, αλλά είναι και αρκετά ευέλικτη ώστε να μπορεί να στηρίξει όλες τις εθνικές νομοθεσίες. Προσαρμόζεται με βάση την αρχή της επικουρικότητας πώς μέσω της εδαφικότητας. Και θα σας το εξηγήσω αυτό σε λίγο. Η γνώμη μου είναι για τα πνευματικά δικαιώματα ότι πρόκειται για ένα δικαίωμα που είναι προσαρμοσμένο στην αγορά, επαρκώς ευέλικτο και ε, το οποίο ε, ο ευρύς χαρακτήρας επιτρέπει να γίνεται άμεσα η προσαρμογή του στη διαρκή καινοτομία που διαπιστώνουμε στο πλαίσιο της ψηφιακής εξέλιξης, της τεχνολογικής εξέλιξης και της πρόοδου της αγοράς. Γιατί τα κείμενα ποτέ δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν την ταχύτητα της εξέλιξης της τεχνολογίας. Πάντοτε θα υπάρχει μια καθυστέρηση ανάμεσα στην εξέλιξη της τεχνολογίας και την εφαρμογή του νόμου. Πέρα λοιπόν από την σταθερότητα των κειμένων, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ώστε οι φορείς στην αγορά να μπορούν να ε, βασιστούν σε αυτό και να το κατανοήσουν, ε, πιστεύω λοιπόν ότι τα πνευματικά δικαιώματα είναι προσαρμοσμένα στην αγορά και από τη στιγμή που υπάρχουν ε, συγγές ή αμφισημίες στα νομοθετικά διδάγματα, μην ξεχνάμε πως έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο γι' αυτό υπάρχει για να συμπληρώσει, για να ερμηνεύσει αυτές τις ενδεχόμενες αμφιβολίες, σημείες που θα λάβει υπόψη ποια είναι τα ήθη και τα έθιμα οι συνήθειες αλλά και πώς θα ερμηνεύσει το κείμενα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει έλλειψη ισορροπίας όπως είπαν ε, ε, οι προλαλήσαντες αλλά πρόκειται για δικαιώματα ευέλικτα ε, και συμπαγή που μπορούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των καταναλωτών. Η αρχή τώρα της εδαφικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε πως οι άδειες εκμετάλλευσης των ε, ε, ταινιών δίνονταν ανά περιοχή, ένα έδαφος. Είναι εδαφικά δικαιώματα δηλαδή και έχει υπάρξει ο ισχυρισμό ότι αυτό, ε, αυτός ο εδαφικός χαρακτήρας εμποδίζει την λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, καμία νομοθετική ευρωπαϊκή διάταξη δεν εμποδίζει τις πολυεδαφικές άδειες εκμετάλλευσης. Δεύτερη διαπίστωση, η δημιουργή σεναρίστες, σκηνοθέτες κτλ. Ε, οι ηθοποιοί και οι ε, διευκολύνουν την κυκλοφορία του περιεχομένου, εκχωρώντας στους παραγωγούς ε, τα δικαιώματα για ολόκληρο τον κόσμο και για ολόκληρη τη διάρκεια της ισχύω αυτών των δικαιωμάτων. Εξ αρχής δηλαδή καθορίζεται αυτό. Τρίτη διαπίστωση, οι πολιτιστικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες της εθνικής ζήτησης περιορίζουν όλα αυτά στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Ε, η πρώτη διαπίστωση, ο πρώτο, το πρώτος λόγος στον οποίο αυτό οφείλεται είναι διότι γνωρίζουμε πως η ε, πολυμορφία, η πολιτιστική, αποτελεί τον πλούτο της Ευρώπης. Ταυτόχρονα όμως η Κομισιόν διαπιστώνει πως τελικά αυτή η πολιτιστική, ε, πολιτιστικός πλούτος παρεμποδίζει τις πολυεδαφικές άδειε εκμετάλλευσης. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε όμως τους καταναλωτές. Ίσως οι καταναλωτές που να ανταποκρίθηκαν να είναι αυτοί που είναι κάπως πιο διεθνείς ε, εγώ σκέφτηκα διάφορα γαλλικά παραδείγματα, γιατί δεν γνωρίζω πολύ καλά τι γίνεται στις υπόλοιπες ε, ευρωπαϊκές χώρες και ποια είναι τα έργα που γνωρίζουν επιτυχία. Πάντως στη Γαλλία το να ζητήσει κανείς να ζητήσει ε, μια πολυεδαφική άδεια εκμετάλλευση για το έργο Plus Belle μου φαίνεται ότι θα ήταν περίεργο και παράξενο γιατί όλο το φιλμ βασίζεται στη Μασαλία, εκτελήσεται στη Μασαλία, ανταποκρίνεται δηλαδή στην γαλλική ιδιαιτερότητα και, και γλώσσα, ώστε τελικά ε, να μην υπάρχουν πολλές ε, εδαφικές αιτήσει για άδειε εκμετάλλευση και όταν αυτές υπάρχουν γίνονται για χώρες που έχουν κοινή, ε, κοινό πολιτισμό ή κοινή γλώσσα. Η σχεδόν πλήρη απουσία λοιπόν πανευρωπαϊκών αδειών προκύπτει από τις πολιτιστικέ ιδιαιτερότητε κάθε κρατου μέλου. Τρέταρτη διαπίστωση. Αποκλειστικότητα είναι το αντιστάθμισμα της προχρηματοδότησης και της χρηματοδότησης της παραγωγής ενός έργου. Είναι απαραίτητη. Ο κατακαιρματισμός λοιπόν της ε, επικράτειας σε εδάφη απορρέει από αυτήν ε, την αποκλειστικότητα. Και είναι απαραίτητη αυτή η αποκλειστικότητα η εδαφική, γιατί είναι η αντιστάθμιση στην προχρηματοδότηση, προχρηματοδότηση ή χρηματοδότηση. Στον μουσικό τομέα, όπου ισχύουν οι πολυεδαφικές άδειε, ένας μέσος προπολογισμό είναι πολύ πιο χαμηλός από ότι ο προπολογισμό μιας ταινία του σινεμά. Μπορεί για κάποιους πολύ γνωστούς ε, καλλιτέχνες να φτάσουμε σε μεγάλους προπολογισμούς. Αλλά ας πούμε μέσος όρος ε, για ένα επεισόδιο ενός σύριαλ στη Γαλλία είναι 710 ευρώ το κόστος για 52 λεπτά. Δηλαδή άμα σκεφτείτε ότι σε ένα σύριαλ μπορεί να φτιάξει κανείς 6-8 επεισόδια θα φτάσει σε ένα κόστος συνολικό 5 εκατομμυρίων ευρώ. Για μία ταινία Μάλλον, τα 5 εκατομμύρια για το Σύριελ θα χρηματοδοτηθούν από, κατά 70% από τους εθνικούς διανομής, γιατί αυτοί έχουν μεγάλη ακροαματικότητα ε, και μάλιστα θα θέλουν αυτοί το πρόγραμμα να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Αυτές οι πολιτιστικές ιδιαιτερότητες λοιπόν μετά για να μπορέσει να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο στην ενιαία αγορά θα είναι εμπόδιο. Θα μειωθεί δηλαδή η ζήτηση. Το 3,8% για ένα σύριλ είναι το κομμάτι των ξένων επενδύσεων. Συν παραγωγή ξένη όταν γίνεται, ε, φτάνει μέχρι 3,8 του προπολογισμού. Θα ζητήσει λοιπόν και εκεί εκείνος αποκλειστικότητα για τα εδάφη που τον ενδιαφέρουν αντίστοιχα με τις πολιτιστικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες. Και έτσι οργανώνεται αυτή η ζήτηση για εδαφικές άδειες εκμετάλλευσης και όχι πολυεδαφικές. Για το σινεμά, ε, μια ταινία κοστίζει γύρω στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ είναι στοιχεία για το 2013. 28,8% το χρηματοδοτεί ο παραγωγός, 24% η εθνική διανομής και 22,5% είναι οι ξένες επενδύσεις. Οι ξένοι λοιπόν επενδυτές θα διανύμουν τις ταινίε αυτές με, με βάση την αξία τους και πώς θα τις αξιολογήσουν σε, με βάση το γούστο των καταναλωτών, τη ζήτηση των καταναλωτών και όπως σας είπα και πριν από λίγο, σπανίως και εγώ θα ζητήσω να δω ένα αγγλικό σύριαλ. Θα δω περισσότερο αυτά που αντιστοιχούν στη δική μου κουλτούρα. Άρα λοιπόν αυτή η ρήτρα αποκλειστικότητα αποτελεί την ε, αμοιβή του επενδυτή στην ουσία. Και αυτή η σύγχυση είναι απαραίτητη. Είναι ε, ε, εκ των για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα και να υπάρξει η δημιουργία σε αυτή τη βιομηχανία. Πέμπτη διαπίστωση. Είδαμε λοιπόν ε, πολιτιστική ιδιαιτερότητα, ε, σπάνια ζήτηση που εξηγείται όμως και από έναν τρίτο παράγοντα, ότι δηλαδή στην εσωτερική αγορά δεν έχουμε πανευρωπαϊκό διανομέα. Δεν υπάρχει κάποιος ευρωπαϊκός διανομέας που να μπορεί οικονομικά να αγοράσει για ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια τα δικαιώματα για να διανύμει τις ταινίες. Η μόνη πανευρωπαϊκή ε, διανομή είναι η γνωστή GAFA, Google, Amazon, ε, Facebook και Apple. Αυτοί έχουν ε, τα μέσα, έχουν τα λεφτά για να το κάνουν. Τι συμβαίνει λοιπόν, Η Ευρωπαίοι παραγωγοί πάνε, μάλλον τελικά αποφασίζουν σιγά σιγά και αυτό ήδη ξεκινάει, το είδαμε για γαλλικές περιπτώσεις, μια, ένα μεγάλο όμιλο κινηματογραφικών παραγωγών που αποφάσισαν να παράγουν με τη Συμφωνία των Δημιουργών να παράγουν προγράμματα που να έχουν πιο διεθνή έτσι, απήχηση. Γιατί? Γιατί αυτά τα αγοράζουν αυτοί οι παγκόσμιοι φορείς. Και εδώ διαπιστώνουμε ακόμη κάτι, με άλλο ένα διακύβευμα και είναι η πολιτική της ε, τιμολόγησης, γιατί βλέπουμε ότι όλη αυτή η οργάνωση της εδαφικότητας βασίζεται σε οικονομικό δικαίωμα και όχι πνευματικό δικαίωμα. Αυτό δεν εμποδίζει σε τίποτα το πνευματικό δικαίωμα της πολυεδαφικές ε, άδειε εκμετάλλευσης. Έχουμε όμως ιδιαιτερότητες πολιτιστικές που αντιστοιχούν στον πλούτο της Ευρώπης και δεν έχουμε και τα χρήματα για έναν πανευρωπαϊκό φορέα ώστε να μπορέσει αυτός να ε, χρηματοδοτήσει και να αγοράσει τέτοιου είδους πανευρωπαϊκές άδειες θα έπρεπε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα ε, μιας εξαίρεσης σε σχέση με το δίκαιο του ανταγωνισμού, ώστε να ε, ε, δημιουργηθεί ένας τέτοιος όμιλος πανευρωπαϊκός για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Η κατάσταση πάντως αυτή δεν εξαρτάται καθόλου στο ελάχιστο από τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά από οικονομικούς παράγοντες. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, διάβασα στον τύπο ότι η Netflix αντιπροσωπεύει το 48,3 ε, εκατομμύρια κόσμο ε, συνδρομητές στον κόσμο. Ενώ το μεγαλύτερο γαλλικό αντίστοιχο συνδρομητικό κανάλι 300.000 κόσμο έχει συνδρομητές. Πώς θέλετε να προτείνει τα ίδια προγράμματα. Θα προτείνει μόνο αυτά που ζητούν οι συνδρομητές του. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να συγχαίουμε την προσβασιμότητα, την κινητικότητα και την ε, διαλειτουργικότητα. Δηλαδή όλα παντού και σε οποιοδήποτε μέσο. Ο κόσμος θέλει να έχει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο που επιθυμεί. Όλοι θέλουν να έχουν λοιπόν πρόσβαση σε όλα, παντού εδώ όπως σας είπα επιμένω είναι οικονομικοί παράγοντες που το εμποδίζουν και όχι ε, τα δικαιώματα τα πνευματικά. Είχαμε ένα πολύ ε, θετικό παράδειγμα όπου η ομάδα εργασίας για το License for Europe ε, ε όπου αποφασίστηκε να συνεργαστούν οι δικαιούχοι όσον αφορά την διαλειτουργικότητα, την, συγγνώμη, την κινητικότητα της προσφοράς και της ζήτησης on demand, το video on demand αυτής της υπηρεσίας και η διαλειτουργικότητα εξαρτάται από τους κατασκευαστές ε, κινητών τηλεφώνων, ε, ε, smartphone, ταμπλέτας κτλ. Όλοι εδώ είμαστε καταναλωτές, όλοι θέλουμε να έχουμε τα πάντα παντού δωρεάν ή εν πάση περιπτώσει όσο γίνεται φθηνότερα, αλλά δεν μπορούμε να ε, καταπατήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό δικαίωμα, το πνευματικό δικαίωμα. Το πνευματικό δικαίωμα λοιπόν είναι απαραίτητο Το δικαίωμα αναπαραγωγής είναι πολύ ε, σημαντικό. Όμως επικρατεί ανισότητα ε, μεταχείρισης ανάμεσα στους ε, μουσικούς, ε, τους ερμηνευτές μουσικούς καλλιτέχνες και τα οπτικοακουστικά μέσα. Η Κομισιόν έπρεπε να κάνει μια μελέτη αντικτύπου που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από τον Ιανουάριο του 2012 και νομίζω προς το, προς το συμφέρον όλων θα ήταν καλό να γίνει αυτή η μελέτη, να εκπονηθεί γιατί η παράταση και η εναρμόνιση της διάρκειας των πνευματικών δικαιωμάτων ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες καλλιτεχνών και δημιουργών θα έχει το πλεονέκτημα να διευκολύνει τις εταιρείε συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων. Τώρα, στην οδηγία του 2001-29 υπάρχει πλήρης κατάλογος των πνευματικών δικαιωμάτων και θα επανέλθω στο θέμα της αμοιβή. Αμοιβή των καλλιτεχνών ερμηνευτών είναι δεδομένου του εύρου τη εκμετάλλευση και των νέων φορέων στην ψηφιακή αγορά, η αμοιβή του θα πρέπει να αυξηθεί. Αυτό είναι βέβαιο και αξίζουν να αυξηθεί γιατί δεν υπάρχει λόγος όταν υπάρχει εκμετάλλευση ενός ε, οπτικού ή μουσικού έργου ε, ε, γίνεται γιατί να μην αμείβεται ο δημιουργός του. Υπάρχει πολύ έντονη ζήτηση των καλλιτεχνών, ερμηνευτών και δημιουργών για μια αμοιβή που θα είναι το δικαίωμα στην αμοιβή remuneration right και που θα επέτρεπε επιπλέον αμοιβή από αυτή που προβλέπεται από την σύμβαση αντίστοιχη με τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και αυτό το προτείνει η ΕΣΑ, ο, Διεθνής, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημιουργών που συγκέντρωσε τις εταιρείε διαχείρισης των δικαιωμάτων, τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιθοποιών... πολύ ε, αντιπροσωπευτικοί δηλαδή οργανισμοί που ζητούν επιπλέον αμοιβή, ένα απαράβατο δικαίωμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να εκχωρήσει που θα είναι ανάλογο με τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης τα κέρδη από την εκμετάλλευση και θα εμπνευστεί ε, από δύο μηχανισμούς δηλαδή την ε, οδηγία 92% που λέει ότι ακόμα κι αν ένας δημιουργός έχει εκχωρήσει τα δικαιώματά του στον παραγωγό, Είτε λοιπόν θα την διαχειρίζονταν συλλογικά, είτε για άλλους θα καταβαλόταν από τον παραγωγό, τον δικαιούχο δηλαδή της άδειας εκμετάλλευσης. Και επιπλέον υπάρχει και άλλη μια πρόταση που προτείνεται από την ΣΑΣΕΜΑ και θα την παρουσιάσει η ΣΑΣΕΜ και είναι μια αντιστάθμιση, αποζημίωση για μια βλάβη που υπόκειται λόγω της αξίας την οποία ε, παίρνουν οι ενδιάμεση ε, για το συγκεκριμένο έργο ή δημιουργία. Αυτό είναι σημαντικό για τον μουσικό τομέα αλλά και για τον οπτικοακουστικό τομέα και γι' αυτό θεώρησα καλό να αναφέρω αυτές τις τέσσερις προτάσεις γιατί έχουμε ε, τρεις Ευρωπαίους ε, ε, φορείς και έναν γαλλικό φορέα για την επιπλέον αμοιβή των καλλιτεχνών και ερμηνευτών. Αυτό το δικαίωμα στην αμοιβή θα απαιτούσαν μια μικρή μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων και όσον αφορά τους καλλιτέχνες ε, ερμηνευτές, αν κάνουμε πολύ εκτεταμένη ερμηνεία της ε, οδηγίας 206-116, ε, εδώ λέμε για... Μιλάμε για μια οδηγία του 92, όπου η ψηφιακή αγορά δεν υπήρχε. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη με εκτεταμένη όπως είπα ερμηνεία ότι εδώ μπορούμε να μιλάμε και για άειλα αντικείμενα, δεν θα χρειαζόταν να μεταρρυθμίσουμε την οδηγία 2001-29 είναι ένα θέμα στο οποίο φυσικά θα πρέπει να εμβαθύνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει το συμπέρασμα είναι ότι το πνευματικό δικαίωμα δεν αποτελεί εμπόδιο στην διασυνοριακή πρόσβαση, δεν αποτελεί εμπόδιο ε, στην κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών. Αντίθετα, θα πρέπει να, η λύση να βρεθεί στο οικονομικό πλαίσιο, μήπω θα έπρεπε να αφήσουμε την αγορά να αυτορυθμιστεί, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, για να δούμε πώ όλοι αυτοί οι φορεί θα τοποθετηθούν, πώ θα προσαρμοστούν, αντί να ανοίξουμε τα πάντα, να αναθεωρήσουμε τα πάντα και να καταστήσουμε αυτό το θεμελιώδε δικαίωμα πιο εύθραυτο, πιο ευάλωτο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου. Επόμενο ομιλητή είναι ο Ζωάν Νοέλ Τρόγκ Γενικός ε, Διευθυντής της ε, Ένωσης των ε, Δημιουργών, Συνθετών και Εκδοτών Μουσικής <clears throat> για τα επόμενα 20 λεπτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πρώτα πάρα πολύ για την οργάνωση αυτού του πάνελ και αυτής της ακόασης. Θέλω να υπογραμμίσω, όπως είπε και η κυρία Κώστα, ότι στον τίτλο αυτού του αυτής της εκδήλωσης μπορούμε να δούμε και την συνωνυμία σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του δημιουργικού τομέα στην Ευρώπη. Θα βασιστώ λοιπόν μονάχα σε ε, πραγματικά γεγονότα γιατί είναι το μόνο σημείο στο οποίο θα συμφωνήσω με τον κύριο Τεμπούς που λέει ότι όλα αυτά που λέμε πρέπει να βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Θα περάσω τώρα στα γαλλικά. Ένα μικρό εισαγωγικό σχόλιο. Μιλάμε εδώ για το copyright. Αυτό θα έπρεπε να το λέμε τα δικαιώματα των δημιουργών και το copyright. Γιατί 26 από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρώπης ζουν σε ένα πλαίσιο δικαιωμάτων του δημιουργού και δύο μονάχα σε ένα περιβάλλον copyright. Θα ήθελα λοιπόν να επιμείνω <clears throat> ότι ιδιαίτερα εδώ στις Βρυξέλλες κάθε φορά που λέμε για το copyright θα πρέπει να μιλάμε και για τα δικαιώματα των δημιουργών και όχι μονάχα για το copyright. Επειδή λοιπόν μιλάμε για, για πραγματικά γεγονότα, είδατε πως μπερδεύομαι με τις κακές συνήθειες της γλώσσα μου, Έχουμε ένα ιδιαίτερο οικονομικό υπόδειγμα που είναι αυτό της συλλογικής διαχείρισης που είναι <clears throat> μια πτυχή της ευρωπαϊκής δημιουργικής και καλλιτεχνικής βιομηχανίας. Όπως είπε ο κύριος Κρέτσμερ στην αρχή, μια από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε είναι το γεγονός ότι γενικά δεν υπάρχει γνώση Ακόμα και εμείς οι ίδιοι στον τομέα του πολιτισμού δεν ξέρουμε ποιο είναι το οικονομικό υπόδειγμα το οποίο επικρατεί στον τομέα του πολιτισμού. Κάποια σχόλια λοιπόν στο σημείο αυτό. Τρία πράγματα θέλω να υπογραμμίσω. Μία εταιρεία όπως η ΣΑΣΕΜ, η Ένωση των Δημιουργών Συνθετών και Εκδοτών Μουσικής που δημιουργήθηκε το 1961 είναι μη κερδοσκοπική ιδιωτικού δικαίου οργάνωση. Είναι τμήμα λοιπόν της οικονομίας της κοινωνικής, της, κοινωνικής, της οικονομίας της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι περίπου 10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όπως υπενθύμησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο στο έγγραφο που τονίζει τη σημασία της κοινωνικής οικονομίας και εδώ σας λέω τι λέει το κείμενο οι κοινωνικές επιχειρήσεις βασίζονται σε προσωπική εμπλοκή των μελών τους στη διαχείριση της εταιρεία και δεν ενδιαφέρονται για την κερδοφορία. Στη δική μου περίπτωση στη ΣΑΣΕΜ το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από δημιουργούς και ε, συνθέτες και από επιχειρηματίες που είναι οι εκδότες το Συμβούλιο αυτό είναι ένα αυτοδιαχειριζόμενο σύνολο, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Όταν μιλάμε λοιπόν για τα δικαιώματα των δημιουργών και το κοπηρά δεν πρέπει να ξεχάσουμε αυτό <clears throat> το γεγονός ότι έχουμε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη που παίζει ακριβώς αυτό το ρόλο. Επίσης, μια εταιρεία όπως η ΣΑΣΕΜ και δεν είναι μόνη, αυτή έχει περίπου 80 ε, 18.000 ε, ε, μέλη συνολικά, 4.000 μέλη κάθε, κάθε χρόνο. Όλοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Creative Commons, δηλαδή τον τρόπο αυτό με τον οποίο μπορούν να φέρουν τα έργα τους για να διαδοθούν στο διαδίκτυο χωρίς καμία αμοιβή. Από τα έργα τα οποία παρουσιάστηκαν λοιπόν, περίπου τα 700 περνούν μέσα από το Creative Commons. Γιατί αυτό, διότι το 2014, όπως ε, πριν από ένα αιώνα κιόλας, πρέπει οι δημιουργοί να ζήσουν από την ε, δημιουργία τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να διατηρηθεί αυτός ο καλλιτεχνικός τομέας. Το ίντερνετ έριξε τους φραγμούς για την παγκόσμια διανομή των έργων και έλυσε ένα σημαντικό πρόβλημα για τους δημιουργούς το 2014 περισσότερο από ποτέ τίθεται όμως το θέμα το πώς θα πρέπει να γίνει η σωστή αμοιβή των δημιουργών. Και εκεί πρέπει να είναι η εστίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τρίτο στοιχείο το οποίο θέλω απλώς να σας δώσω. Μια ένωση όπως η δική μας πέρσι διένυμε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε 300.000 περίπου δημιουργούς συνθέτες και εκδότες στον κόσμο. Επειδή πολλές φορές υπάρχει το σύστημα αμοιβαίας εκπροσώπησης στις επιχειρήσεις, ένα αποτελεσματικό σύστημα, όπως αυτό που γίνεται με το roaming στην κινητή τηλεφωνία, επιτρέπεται με τον τρόπο αυτό ο κάθε καλλιτεχνικός δημιουργός να έχει άδειες με ένα απλό τρόπο για την εκμετάλλευση των έργων. Το ένα δεύτερο σχόλιο σε σχέση με αυτό το ποσό είναι ένα παγκόσμιο σύστημα και είναι ένα σύστημα το οποίο έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά και με διαφάνεια, αλλά κυρίως ένα σύστημα το οποίο εξασφαλίζει την αλληλεγγύη. Σε μια εταιρεία δημιουργών, όταν εγώ παίρνω μια άδεια για τα μέλη μου, όπως οποιοδήποτε άλλος επικεφαλής μια συλλογικής ε, οργάνωσης, μπορώ να διαπραγματευτώ με το YouTube, με το Netflix για όλα τα μέλη μου. Τα εφαρμόσω λοιπόν αυτά στις μεγάλες εταιρείες και τα εφαρμόζω και στους πιο μικρούς από τους παραγωγούς μας και τους συνθέτες. Χάρη σε αυτήν την αμοιβή του έργου τους μπορούν να επιβιώσουν. Από τα 4.000 μέλη που είχαμε πέρσι, που προσθέθηκαν πέρσι, το μεγαλύτερο μέρος δεν ζουν από την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα και φυσικά πρέπει να γνωρίζετε εσείς πώς θα πρέπει να εξασφαλιστεί η διατήρηση αυτού του αποτελεσματικού μοντέλου που επιτρέπει σήμερα στην Ευρώπη σε περίπου ένα εκατομμύριο δημιουργών κάθε είδους να έχουν την ελπίδα να ζήσουν από το έργο τους <clears throat> χωρίς πολλές πολυτέλειες, αλλά είναι ένα δικαίωμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το διατηρήσουμε. Έρχομαι τώρα στο πιο οικονομικό τμήμα της παρουσίασης. Αν πάρετε τον καλλιτεχνικό και δημιουργικό τομέα, τον πολιτιστικό τομέα, Στη Γαλλία πέρσι έγινε μια μελέτη την οποία μπορώ να σας παρουσιάσω. Ξέρω ότι και μια αντίστοιχη μελέτη μπορεί να σας δοθεί σε τις εβδομάδες στις 2 Δεκεμβρίου. Θα σας δώσω λοιπόν κάποια στοιχεία και μπορείτε με τον τρόπο αυτό να καταμετρήσετε το οικονομικό βάρος αυτού του τομέα στην Ευρώπη. Σας υπενθυμίζω ότι όλες οι εργασίες που θα πρέπει να κάνετε εσεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλες οι αποφάσεις που θα πρέπει να λάβετε θα έχουν άμεσο αντίκτυπο θετικό ή αρνητικό σε σχέση με τη χρηματοδότηση αυτού του τομέα. Πρώτο δίδαγμα λοιπόν, στον τομέα αυτό υπάρχει μια πολυμορφία για τις ε, οικαστικές τέχνες είναι μια από τις σημαντικότερες από τους κλάδους στην Ευρώπη. Η γλυπτική, η ζωγραφική, η φωτογραφία υπάρχουν ορισμένοι τομεί οι οποίοι είναι πολύ συγκεντρωμένοι, άλλοι είναι αποκεντρωμένοι. Δεν έχει σημασία όμω. Αν πάρετε το παράδειγμα τη Γαλλική και μόνο αγοράς, ο τομέα αυτό είναι ο τρίτο τομέα σε απασχόληση και είναι ένα τομέα ο οποίο έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρο από την ε, βιομηχανία του αυτοκινήτου, περισσότερο από τα αγαθά πολυτελεία και τα αμυντικά θέματα. Είναι ένα τομέα ο οποίο στη Γαλλία περιλαμβάνει θέσεις εργασίας οι οποίες δεν μπορούν να μετακινηθούν. Όταν έχουμε πάνω από 10% ανέργων και πάνω από 25% των νέων είναι άργοι, για μένα ένα από το σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε την απασχόληση σε τομείς οι οποίοι έχουν δυνατότητα ε, ανάπτυξης. Και θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Ένα τρίτο δίδαγμα, αν δούμε αυτό το τομέα, βλέπουμε την τεράστια πολυμορφία που υπάρχει σε ό,τι αφορά τα υποδήματά του. Ορισμένα κομμάτια είναι μη κερδοσκοπικά, όπως η εταιρεία Musecam, άλλα είναι ε, μοντέλα κερδοσκοπικά και άλλα είναι μοντέλα δημόσιας χρηματοδότησης. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς, όπως βλέπετε και σε αυτό τον ε, πίνακα, ο τομέας της εκπαίδευσης, ο τομέας της υγείας, όπου υπάρχει επικάλυψη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων ένα σημαντικό τώρα δίδαγμα για την ευρωπαϊκή μελέτη η οποία θα σας δοθεί στις 2 Δεκεμβρίου είναι απαραίτητο να καταλάβετε ότι είναι αυτή αναπτυσσόμενη τομής. Το κύριο δίδαγμα της μελέτης αυτής, η οποία είναι μια ανεξάρτητη μελέτη, έγινε επί τη βάση μιας διαδικασίας ε, δημόσιου διαγωνισμού και εξάλλου είναι και μια συντηρητική μελέτη γιατί μετράει μονάχα το συνολικό ε, τζίρο και όχι μονάχα την προσθέμενη αξία. Λοιπόν, δεν λαμβάνει υπόψη την πλήρη προσθέμενη αξία. Στον τομέα της μουσικής πήραμε τον ε, κύκλο εργασιών των ε, καλλιτεχνικών δημιουργών, των ε, κατασκευαστών μουσικών οργάνων, των δασκάλων της μουσικής, των ε, δισκογραφικών εταιριών, των δισκοτέκ, των ραδιοφώνων, των φεστιβάλ μουσικής κτλ. που μεταλαμβαδεύουν τη μουσική δημιουργία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταμετρήσουμε την αξία αυτού του τομέα. Αν υπάρχει λοιπόν ένα ενδιαφέρον δίδαγμα, είναι ότι αν πάτε την πιο δύσκολη εποχή της κρίσης, 2008-2012, η μέση τάση της απασχόλησης στην Ευρώπη ήταν μείον 0,7% το χρόνο για τον πολιτιστικό τομέα και το δημιουργικό τομέα μεταξύ του 2008 και 2012 ήταν ακριβώς το αντίθετο. Συν 0,7% αύξηση το χρόνο. Αυτό είναι το πρώτο ενδιαφέρον λοιπόν μήνυμα. Ένα δεύτερο μήνυμα, η ευρωπαϊκή μελέτη που θα σας δοθεί θα επιβεβαιώσει τη στατιστική που βλέπουμε στην Γαλλία, σε μία από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η πολιτιστική και δημιουργική, ο δημιουργικός κλάδος είναι ο τρίτος σε αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν τίθεται λοιπόν το θέμα της ανάπτυξης των δικαιωμάτων των ε, δημιουργών και του copyright στην Ευρώπη, ειλικρινά μπορούν να υπάρχουν πάρα πολλά τεχνικά θέματα, τα οποία έχουν τη σημασία τους και πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια. Αλλά όλα αυτά πολλές φορές είναι θέματα λεπτομέρειες σε σχέση με το ουσιαστικό ερώτημα που είναι πώς θα μπορέσουμε μέσα από τα δικαιώματα των δημιουργών και το copyright μπορείτε να συμβάλλετε στην ανάπτυξη αυτού του τομέα. Μήπως υπάρχει κάποια ελπίδα ότι μετά από πέντε χρόνια όταν τελειώνει η θητεία αυτού του ε, κοινοβουλίου θα έχει φτάσει στα 10 εκατομμύρια θέσεων απασχόλησης και όχι 7 όπως τώρα. Και αντίθετα τα λόμπι τα οποία σας προτείνουν συνέχεια να υπάρξει απομείωση των δικαιωμάτων προστασίας αυτά τα λόμπι που ανέφεραν ορισμένοι και τα οποία είναι όλα σχεδόν έξω από την Ευρώπη. Μήπως είναι σε θέση αυτά τα λόμπι να δημιουργήσουν εκατομμύρια θέσεις εργασία στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα λοιπόν το οποίο πιστεύω πρέπει να θέσουμε και αυτό συμπεριλαμβάνει και τους τομείς όπου το δικό σας κοινοβούλιο θα πρέπει να φέρει και ενωτόμες λύσεις και θα έρθω στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασής μου. Θα ήθελα παρόλα αυτά ναι, ξέχασα να σας ε, πω ότι εδώ στην οθόνη βλέπετε τη σύνοψη αυτής της μελέτης, η οποία σίγουρα θα είναι σύντομα δημόσια. Προτού περάσω σε μια πιο νομικού χαρακτήρα πρόταση σε σχέση με την μεταφορά αξίας, θα ήθελα να σας τονίσω ότι ο τομέας αυτός είναι ένα οικοσύστημα το οποίο έχει συνοχή. Στον τομέα αυτό η δημόσια χρηματοδότηση και η ιδιωτική χρηματοδότηση λειτουργούν αρκετά συμπληρωματικά. Ένα τρίτο στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι παντού στην Ευρώπη η δημόσια χρηματοδότηση του πολιτισμού και της, του δημιουργικού κλάθους είναι λιγότερο από 10% του συνόλου. Όπως σας έλεγα προηγουμένως, είναι ένας τομέας ο οποίος είναι σε μεγάλο βαθμό βασιζόμενος στην ιδιωτική δυναμική και καθορίζεται η υγεία τους από τη ρύθμιση, είτε είναι η ρύθμιση της προσφοράς, είτε είναι η ρύθμιση δημοσιονομική. Το ενιαίο, η ενιαίο τίμημα για τα βιβλία είναι κάτι το οποίο το οφείλουμε στην Ισπανία που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά. Πρέπει λοιπόν η ρύθμιση να είναι προσαρμοσμένη στι σύγχρονε εποχέ και τι ανάγκε. Παραδείγματο χάρη, το ιδιωτικό αντίγραφο. Αυτό είναι μια γερμανική εφεύρεση. Το ιδιωτικό αντίγραφο είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί σήμερα σε πάνω από 50 χώρε στον κόσμο. Είναι η πρώτη πηγή χρηματοδότηση για την ε, αμοιβή των δημιουργών στο Μπουρκίνα Φάσο ή την Αλγερία. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι αρκετά θετικό γιατί επιτρέπει την ε, σύλληψη της αξίας, την μετάφραση σε χρήματα της αξίας αυτής. Αυτή τη στιγμή η Apple είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα αυτό. Αλλά τα λεφτά της Apple δεν έρχονται από το iTunes ή από το ίντερνετ έρχονται από τα κινητά τηλέφωνα, τα τάμπλετ και τους υπολογιστές που πουλάει και τα πουλάει αρκετά ακριβά. Υπήρξα γενικός διευθυντής ενός ε, φορέα τηλεπικοινωνίας στην ε, Γαλλία. Α, έρχομαι από την άλλη μεριά του φεγγαριού γιατί ήμουνα κομπιουτεράς και έχω δουλέψει στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες. Ένα τηλέφωνο όπως αυτό που κρατάω στα χέρια μου όταν ήμουν επικεφαλιστής Orange στη Γαλλία πριν από 7 χρόνια 6 εκατομμύρια τέτοια πουλάμε το, πουλάγαμε το χρόνο. Αυτό θα μπορούσαμε σήμερα να το πληρώσουμε, να το πουλήσουμε μόνο 40 ευρώ, γιατί δεν έχει μεγάλη αυτονομία, άμα πέσει και σπάσει χαλάει και ως τηλέφωνο είναι πολύ ε, μέτριο. Αλλά γιατί το πληρώνω, γιατί το πουλάω, 15 το αγοράζω σήμερα 15 φορές και χαίρομαι από ότι το αγόραζα τότε όταν ο Ζωάν Μισελ Ζάρ, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος αυτής της εταιρείας, έλεγε ότι το smart, τα smartphones είμαστε εμείς ήδη. Γιατί λοιπόν οι καταναλωτές πληρώνουν τα μάτια της Παναγιάς για να πάρουν αυτό το, το τηλέφωνο. Γιατί αυτό δίνει τη δυνατότητα να έχουν μια πρόσβαση στην ε, καλλιτεχνική παραγωγή. Γι' αυτό θέλω να χαιρετήσω τη θέση του Κοινοβουλίου και θέλω να χαιρετήσω και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δικαίωσε την Αυστρία έναντι του Amazon. Πρέπει λοιπόν να επεκτείνουμε αυτό το σύστημα της αντιγραφής και όχι να το καταργήσουμε. Ας εναρμονίσουμε προς τα πάνω. Όπως είπε ο Ματέο Ρέντσι, ο οποίος είπε να διπλασιαστούν οι φορολογίες για τα iPhone και τα iPad για το ιδιωτικό αντίγραφο. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό που κάνουν και οι Γερμανοί, να υπάρχει ένα ισοδίκαιο ε, σύστημα για την αμοιβή των δημιουργών και δεν οι καταναλωτές οι οποίοι θα πληρώσουν. Οι καταναλωτές λοιπόν για τους καταναλωτές έδειξαν ότι τα προϊόντα πουλούνται πιο ακριβά στις χώρες όπου δεν υπάρχει το ιδιωτικό αντίγραφο. Αυτό το τηλέφωνο πουλιέται πιο ακριβά στο Λονδίνο που δεν υπάρχει το ιδιωτικό αντίγραφο από ότι στη Γαλλία που υπάρχει. Κλείνω λοιπόν αυτό το γενικό ε, σχόλιο. Βλέπετε εδώ πέρα την πολυμορφία του μοντέλου. Θέλω να υπογραμμίσω το εξή. Η μεταφορά της αξίας είναι μια πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε μέσα από τις άδειε και εδώ ο, πρόεδρος, ο πολύ σωστά τόνισε ότι η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι αυτή που θα καθορίσει πώς θα γίνει αυτή η μεταφορά αξίας. Έθεσε νομίζω το σωστό ερώτημα. Και αν πρέπει να αντιμετωπίσετε κάτι, είπε ότι το μοντέλο μας θα πρέπει να είναι το παλαιό, το, το σύστημα της Γερμανίας και όχι το σύστημα του Google. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια λογική η οποία πάλι έλκεται από το γαλλικό σύστημα, αυτό το οποίο ονομάζω εγώ τον ψηφιακό τροχό. Άμα πάρω το συνολικό τζίρο των ψηφιακών βιομηχανιών, του ψηφιακού κλάδου σε όλη τη χώρα, σε ποιο βαθμό οι τομείς αυτοί χρηματοδοτούν την κουλτούρα. Αν δείτε, έχει το τομέα του δικτύου, των συσκευών και του δικτύου. Βλέπετε λοιπόν τους ε, παίκτες και βλέπουμε ότι παρά την ε, επιτυχία του Διζέρ, οι περισσότεροι φορείς για το ίντερνετ και για, τα, για τις συσκευές είναι έξω από την Ευρώπη. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα έχουμε ανεξάρτητες τηλεπικοινωνίες. Αν πάρετε το παράδειγμα της Γαλλίας, το συνολικός τζίρος όλων αυτών το 2012 ήταν 49 δισεκατομμύρια ευρώ. Άμα δείτε ποιο είναι το τμήμα το πράσινο του δικτύου, βλέπετε ότι από διάφορα συστήματα ρύθμισης τα πνευματικά δικαιώματα ή ο φόρος για τους παρόχους υπηρεσιών που ενεκρίθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 33 δισεκατομμύρια συμβάλλουν όλοι αυτοί μόνο με 600 εκατομμύρια. Αν δείτε τις συσκευές από 13 δισεκατομμύρια που παίρνουν αυτοί οι οποίοι εισάγουν τα προϊόντα αυτά τα ηλεκτρονικά στην Ευρώπη και περιλαμβάνει αυτό και το δικαίωμα αμοιβή μέσω των φωτοτυπιών φτάνουμε περίπου 230 εκατομμύρια από τα 13 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ περιορισμένο τμήμα του τζίρου των μεγάλων εταιριών οι οποίοι έρχονται με το lobby Digital Europe και λένε στην Ευρώπη ότι αν μπορούσαμε να εναρμονίσουμε και να άρουμε το ευρωπαϊκό σύστημα για την προστασία των δημιουργών θα είχαμε περισσότερη δημιουργία αξίας. Μα αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Αυτή η αξία κυρίως φεύγει από τη ρύθμιση και βγαίνει και από την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υπηρεσίες ίντερνετ. Μπορούμε να έχουμε αδειοδότηση, αλλά η οδηγία όπως του 2000 όπως έχει δεν δίνει καμία δυνατότητα. Το σκοτεινό τμήμα είναι αυτό το οποίο καλύπτεται από κάποια αμοιβή, ενώ τα υπόλοιπα όχι. Έχουμε λοιπόν μέσα από τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις των Δημιουργών υποβάλλει μια πρόταση η οποία ελπίζουμε ότι θα μπορέσει τους επόμενους μήνες να εξεταστεί από τους Ευρωπαίους νομοθέτες. Το λέμε Internet intermediaries Creative Contribution. Συμβολή στη δημιουργική βιομηχανία των ενδιαμέσων του ίντερνετ. Πώς λοιπόν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι εταιρείε όπως η Google θα συμβάλλουν στον πολιτιστικό και καλλιτεχνικό τομέα. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει ένα το ευρωπαϊκό πλαίσιο και δεν θα σταθώ στα νομικά επιχειρήματα. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την οδηγία του 2000. Εγώ ήμουνα ε, σύμβουλος του Πρωθυπουργού και η Μαρία ήταν μέσα στην ομάδα που ε, εκπώνησε αυτή την οδηγία. Τότε η Ευρώπη ήταν πρωτοπόρος στα κινητά τηλέφωνα ήταν πολύ ισχυρή στην πληροφορική και στα θέματα του ίντερνετ. Τώρα οι τομείς αυτοί έχουν πεθάνει ουσιαστικά στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν εταιρείε, δεν υπάρχει Sinclair, δεν υπάρχει Ericsson, δεν υπάρχει η Siemens για τα κινητά τηλέφωνα. Αλλά έχουμε ακόμα δημιουργικό κλάδο στην Ευρώπη και θα πρέπει ο νομοθέτης να σκεφτεί αυτό και να θέσει εκεί την έμφαση στις αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν με στόχο να ενισχύσει το επίπεδο προστασίας των δημιουργών και επίσης να ενισχύσει το επίπεδο ρύθμισης και με αποτελεσματικό τρόπο ευχαριστώ. Thank you very much for your... Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλια που ακούσαμε. Τελευταίος ομιλητής τώρα είναι ο καθηγητής Μάλτε Στίπερ της έδρας αστικού δικαίου και δικαίου ανταγωνισμού στο Πανεπιστήμιο Μαρτίνου Λουθύρου της Χάλε Βιτεμβέργης και μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για το δίκαιο βιομηχανικής διοκτησίας στην Γερμανία. Τα επόμενα 20 λεπτά μπορείτε να ομιλήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σβόμποτα και εσάς κυρία Κώστα για την διοργάνωση της ακροάσεως σήμερα και μάλιστα σε τόσο πρώιμο στάδιο της νομοθετικής περίοδου. Όπως και ο κύριος Τρόγκ θα ομιλήσω κι εγώ την μητρική μου γλώσσα. Ο κύριος ε, Ντουμπός ανέλησε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία του δικαίου του δημιουργού και τόνισε ότι είναι σημαντικό ότι από τις 10.000 περίπου απόψεις που υποβλήθηκαν από, στην διαβούλευση, πάνω από τις μισές προήρθαν από τελικούς καταναλωτές, από χρήστες δηλαδή. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει το δικαίωμα και το δίκαιο της προστασίας του δημιουργού και για τους ε, τελικούς καταναλωτές. Στον αναλογικό κόσμο, ο καταναλωτής δεν ερχόταν σε επαφή με το δικαίωμα, η τελική χρήση από τον τελικό καταναλωτή, δηλαδή η ακρόαση του ακρόαματος ή η θέαση του θεάματος, γινόταν μόνο έμεσα, μόνο πλήρωνε το βιβλίο ή τον ε, ε, σύμπαγη δίσκο ή πήγαινε στον κινηματογράφο. Η αποζημίωση του δημιουργού δεν γινόταν από τον τελικό χρήστη, αλλά από τους παραγωγούς, εκδότες ή διανομής των ε, ταινιών κινηματογράφου. Έτσι λοιπόν, εκεί έχουν εντοπίσει, εκεί έχουν στοχεύσει ε, τα δικαιώματα, τα ε, δίκαια αυτά. Όμως στην ψηφιακή εποχή τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο ίδιος λοιπόν ο τελικός καταναλωτής γίνεται ο αξιοποιητής του έργου, αυτός που χρησιμοποιεί δηλαδή τελικά το έργο μέσω του διαδικτύου. Ακόμα και η απλή ακρόαση ενός ε, αρχείου μουσικής σε ένα iPod ή ε, FES τηλέφωνο ή ταμπλέτα απαιτεί ολόκληρη σειρά τεχνικών αντιγραφής που σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο τουλάχιστον παρεμβαίνουν στο δικαίωμα του δημιουργού. Η διάκριση που γινόταν προηγούμενα ανάμεσα σε ιδιωτική και δημόσια χρήση δεν λειτουργεί πλέον μέσα στα πλαίσια του Web 2.0 και επιτρέπει και όλα σε ορισμένους την παράνομη χρήση του διαδικτύου από ασφαλή θέση στο εξωτερικό. Μέχρι τώρα το δίκαιο της προστασία του δημιουργού βασιζόταν απλά σε μια αυστηρότερη ρύθμιση, από την οποία όμως εποφελούνταν μονάχα οι μεγάλοι διανομής, οι οποίοι δεν θέλουν να αλλάξει και τίποτα στο ε, δίκαιο προστασία του δημιουργού, κάτι που οδηγεί όμως επιτέλους σε μια υπερτροφία των δικαιωμάτων προστασίας, δηλαδή υπερβολική προστασία, κάτι που καθιστά δύσκολο στον τελικό καταναλωτή να αντιληφθεί για ποιο λόγο χρειάζεται το δίκαιο προστασίας του δημιουργού. Και αυτό είναι πιο επικίνδυνο για το δίκαιο του δημιουργού από ίσως μεμονωμένες παραβιάσεις του δικαίου αυτού. Χρειάζεται λοιπόν ένα σύγχρονο δίκαιο προστασίας του δημιουργού, το οποίο να λάβει υπόψη και τα συμφέροντα της, ε, του κοινού συνόλου για πρόσβαση σε καλλιτεχνικά έργα και βεβαίω και για την προστασία άλλων δημιουργών που θέλουν να έχουν πρόσβαση στο ε, δημιούργημα, στο ε, έργο. Και πρέπει να επιβληθούν και περιορισμοί, χωρίς βεβαίως να λησμονηθούν ή να λησμονηθεί η προστασία των ε, δημιουργών. Έτσι όμως προς το συμφέρον και των δημιουργών και των τελικών καταναλωτών σημαίνει ότι λιγότερο δίκαιο προστασίας είναι καλύτερο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και το πώς μπορεί να γίνει αυτό στο μέλλον θα σας το εξηγήσω φωτίζοντας τρεις πτυχές. Πρώτα, το αντικείμενο προστασίας, δηλαδή ποιο είναι το αντικείμενο που προστατεύεται. Δεύτερο, το εύρος της προστασίας, δηλαδή ποιες χρήσεις μπορεί να απαγορεύσει ενδεχομένως ο κάτοχος του δικαιώματος. Και τρίτο, η πυκνότητα των ρυθμίσεων, δηλαδή ποια νομοθετικά μέτρα πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρώτα για το αντικείμενο της προστασίας. Αντικείμενο της ε, προστασίας, και εδώ βεβαίως συμφωνούν οι περισσότερες ένωμες τάξεις, είναι το έργο ποιες είναι οι απαιτήσει τώρα προς το έργο και επομένως προς το ε, δίκαιο της προστασίας, αυτές είναι πολύ διαφορετικές, ρυθμίζονται πολύ διαφορετικά στις διάφορες ονομές τάξεις. Όμως είναι απαραίτητο να υπάρξει ενιαίος ορισμός του ε, αντικειμένου προστασίας, διότι εν τέλει πρόκειται για μια ενιαία αγορά και δεν θα είναι δυνατή αυτή εάν γίνεται η προστασία σύμφωνα με 28 διαφορετικές ένομες τάξεις. Επομένως, η πρώτη ερώτηση που θα πρέπει να ρυθμίσει ο νομοθέτης στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πρώτα-πρώτα τι σημαίνει έργο. Ποιο είναι λοιπόν το αντικείμενο προστασίας του δικαίου προστασίας. Μέχρι τώρα ο ορισμός γίνεται μονάχα σε ό,τι αφορά τράπεζε δεδομένων, λογισμικά και φωτογραφίες. Δεν μπορεί όμως αυτό να είναι αντιπροσωπευτικό του υποπροστασία έργου. παρόλα αυτά, χρειαζόμαστε και για άλλα έργα, ιδίως για μουσικά έργα, για και κινηματογραφικές ταινίε, για συγγράμματα, χρειαζόμαστε συγκεκριμένο ορισμό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βέβαια από τις υφιστά, ορισμού ορισμούς κατά αναλογία συμπεραίνει ότι το δικαίωμα το δίκαιο προστασίας αναφέρεται μοναχά σε ίδιο πνευματικό έργο, ίδια πνευματική δημιουργία. Όμως αυτό δεν μπορεί να παραμείνει στα χέρια της νομολογίας, θα πρέπει να επεκταθεί και μάλιστα νομοθετικά σε όλες τις μορφές δημιουργίας. Έτσι λοιπόν, εποφελία και δημιουργών και καταναλωτών θα πρέπει να οριστεί ποια είναι η ίδια καλλιτεχνική δημιουργία. Η δημιουργία. Και αυτή δεν μπορεί να μείνει στο κενό διότι δεν είναι δυνατόν να προστατεύεται ως δικαίωμα δημιουργού και η τελευταία απλή φωτογραφία που έχει αναρτήσει κάποιος στο διαδίκτυο. Όχι λοιπόν απλά skill and labor προστασία και προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Όχι λοιπόν απλά μια τεχνική επεξεργασία. Αυτά ζητεί άλλωστε τις αποφάσεις του και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν προστατεύονται λοιπόν ορισμένες μορφές δημιουργίας όπως η απλή συλλογή πληροφοριών. Διότι μόνο με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατόν από πλευράς δικαίου δημιουργού και οι, αυτοί που μεταφέρουν ε, πληροφορίες να αποφασίζουν να αποφασίζει δηλαδή ο τελικός καταναλωτής πώς θα τις χρησιμοποιήσει. Η μορφή που θα, που θα περιβληθούν αυτές οι, οι, ε, πληροφοριών μπορεί να είναι άξια προστασίας. Η απαραίτητη ο απαραίτητος περιορισμός της προστασίας σε αυτές τις ε, πρωτότυπες δημιουργίες δεν μπορεί να επιτρέπει ωστόσο και την εφαρμογή του συγγενούς δικαίου που ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις διότι με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ των ενδιαμέσων πληροφοριών, των ενδιαμέσων δηλαδή που παρέχουν πληροφορίες. Όπως το γερμανικό δίκαιο για τους εκδότες που υποτίθεται ότι απαγορεύει στο Google σε περιπτώσεις έρευνας στο Google να δείχνει αυτό τμήματα από άθα εφημερίδων χωρίς προηγουμένως να έχει χορηγηθεί άδεια από τον εκδότη και επομένως να έχουν καταβληθεί τέλεια από πλευράς Google. Ένα σχετικό νομοθέτημα για ένα τέλος Google έχει εκδώσει και η Ισπανία που θα αρχίσει να ισχύει από τις αρχές του επόμενου χρόνου. Αυτά δεν μπορεί να τα προστατεύσει το δίκαιο προστασίας του δημιουργού. Αυτός ο γερμανικός αλλά και ο ισπανικός τώρα νόμος Google δεν μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση τέτοιου ευρωπαϊκού ορισμού της έννοιας του έργου, του προστατευτέου έργου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάθε δημιουργία λίγο πολύ βασίζεται σε κάποια προϋπάρχοντα στοιχεία ή διασυνδέεται με κάποια που ήδη υπάρχουν. Το γεγονός ότι η δημιουργία μπορεί να σημαίνει και επεξεργασία ενός άλλου ήδη υφιστάμενου έργου δεν ρυθμίζεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και περαιτέρω επεξεργασία λοιπόν και συνδυασμό προϋπαρχόντων έργων όπως Remix και Mashup. Εκεί χρειάζεται ωστόσο εναρμόνιση του δικαίου προστασίας του δημιουργού πανευρωπαϊκή. Η διάδοση δε τέτοιων user-generated content δεν πρέπει να παραβιάζει το δίκαιο του δημιουργού του προϋπάρχοντος έργου, εφόσον δεν επιδιώκονται εμπορικά ωφέλη. Ήδη στην σχετική πράσινη βίβλο του 2008 έχουν ε, περιληφθεί τα σχετικά, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα και είναι απαραίτητο να γίνει εναρμόνιση. Και από την άλλη μεριά θα πρέπει να ρυθμιστεί ρητά ότι τέτοιες επεξεργασίες προϋπαρχόντων έργων, τροποποιήσεις δηλαδή προϋπαρχόντων έργων, από την πλευρά τους είναι πάλι και αυτές άξιες προστασίας, εφόσον σημαίνουν δημιουργική επένδυση, ε, διανοητική επένδυση του ίδιου του δημιουργού τους. Αυτό στις περισσότερες ένομες τάξεις ρυθμίζεται ήδη. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά μεταφράσεις. Αλλά δεν υπάρχει αυτό στο ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι ένα κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Λιγότερα σημαίνουν εν τέλει περισσότερα. Αυτό ισχύει όμως και για το εύρος της προστασίας. Από την άποψη του χρήστου των προστατευόμενων έργων, σημασία έχει πόσο μπορεί να χρησιμοποιήσει τα έργα αυτά χωρίς άδεια του δημιουργού. Όμως το εύρος της προστασίας αφενός ορίζεται από το εύρος των απαγορεύσεων που μπορεί να επιβάλλει ο δημιουργός, από την άλλη μεριά από τους φραγμούς που επιβάλλει το δίκαιο προστασίας του δημιουργού. Για παράδειγμα, παραθέσεις από ξένα έργα ή ε, ιδιωτικά αντίγραφα που ανέφερε προηγουμένως ο κ. Στρόγκ. Εάν τώρα επιτρέπεται μια συγκεκριμένη χρήση ενός έργου, αν δηλαδή ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα έργο χωρίς πρώτα να ζητήσει άδεια του δημιουργού, αυτό προκύπτει από συνολική πρώτα εξέταση αφενός των ενδεχόμενων απαγορεύσεων του δημιουργού, αλλά αφετέρου και των ενδεχόμενων φραγμών που υπάρχουν για τη χρήση του έργου. Εάν το εύρος των απαγορεύσεων έχει μεν εναρμονιστεί από τη σχετική οδηγία, μέχρι τώρα ωστόσο από το δίκαιο της ενώσεως μέχρι τώρα έχουν αρμονιστεί μονάχα δύο φραγμοί. Αφενός η τεχνική απαραίτητη ενδιάμεση αποθήκευση σε υπολογιστές του διαδικτύου και αφετέρου η ρύθμιση πρόσφατα σε οδηγία και ενδεχομένω. τρίτο η εφαρμογή της σύμβασης του Μαρακέσου που ενδέχεται να περιληφθεί στο ενωσιακό δίκαιο. Εξάλλου η οδηγία InfoSoc δεν προβλέπει δεσμευτικά υποχρεωτικούς φραγμούς, αλλά ένα δυνητικό κατάλογο 20 μέτρων που μπορούν να επιβάλλουν χωρισμένοι, αλλά δεν είναι υποχρεωμένες. Θα έλεγε κανείς, φραγμή όλων των χωρών ενωθείτε. για να περιληφθούν στις ένομες τάξεις όλων των χωρών μελών. Αυτό όμως στην ουσία είναι το αντίθετο της εναρμόνισης και αυτό προκαλεί προβλήματα από δυο απόψεις. Αφενός τέτοια επιλεκτική δυνητική ρύθμιση δεν μπορεί να εξασφαλίσει ενιαίο επίπεδο προστασίας στην ενιαία αγορά. Έτσι λοιπόν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Για παράδειγμα κατά πόσο επιτρέπονται παροδίες γνωστών προεπαρχόντων έργων. Οι Γάλλοι είναι πολύ γενναιόδοροι, οι Γερμανοί είναι μάλλον περιοριστικοί. Πάντως, το όποιος βάλει τέτοια παροδία έργου στο διαδίκτυο, σε ορισμένες περιπτώσεις παραβιάζει το, δικαίο, το δίκαιο προστασίας του δημιουργού, σε άλλες χώρες όχι. Υπάρχει λοιπόν μια σημαντική απόκληση δικαίου προστασίας. Και βέβαια υπάρχουν αποκλήσεις του δικαίου που θα πρέπει να ξεπεραστούν. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ζητήσει να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση της έννοιας της παροδίας. Αλλά βεβαίω οι χώρες μέλη μπορούν ακόμα να απαγορεύσουν απολύτως τις παροδίες και αυτό είναι, είναι, είναι δυνατόν να γίνει ακόμη. Μπορούν οι χώρες μέλη επίσης να προβλέψουν περισσότερους φραγμούς. Αυτό όμως δεν μπορεί να το επιτρέψει ο Ευρωπαίος νομοθετής. Πρέπει να εναρμονιστούν και οι φραγμοί που προβλέπουν διάφορες ένομες τάξεις για να εξασφαλιστεί η μεταχείριση δημιουργών και καταναλωτών. Από την άλλη μεριά, εξαντλητικός κατάλογος των δυνητικών φραγμών θα ήταν υπερβολικά άκαμπτος και δεν θα επέτρεπε να τα αποκρίνονται ένομες τάξεις σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις, για παράδειγμα η αναζήτηση εικόνων στο διαδίκτυο. Τα λεγόμενα thumbnails δηλαδή, τα οποία επιτρέπονται στο διαδίκτυο. Άλλωστε ο δημιουργός δεν έχει κανένα συμφέρον να τα απαγορεύσει αυτά, με τα μικρά εικονίδια δηλαδή τα οποία ε, δίνουν μια ιδέα για το ποια θα είναι η τελική εικόνα που θα μπορούσε να κατεβάσει από το διαδίκτυο. Εδώ πρέπει επίσης να γίνει ε, ρύθμιση. Το ίδιο προβληματικές είναι οι ρυθμίσεις φραγμών που ε, επιτρέπουν μοναχά αναλογική χρήση. Σε πολλούς τομείς η ψηφιακή τεχνολογία έχει παραγωνίσει τις παλιές αναλογικές χρήσεις. Για παράδειγμα, για την χρήση ε, εγχειριδίων που κατεβάζουν από το διαδίκτυο για τη διδασκαλία σε ε, πανεπιστήμια. Ποιος κάνει τώρα course pack, όπως λέγονται αυτά, σε χαρτί. Αυτή η απολύθωση του ευρωπαϊκού δικαίου σε συγκεκριμένες μορφές χρήσης που τεχνικά είναι ξεπερασμένες πρέπει να απαγορευτεί. Ο στόχος αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα με ενδεικτικές απαριθμίσεις και με διατυπώσεις που να αφήνουν άνοιγμα στις τεχνολογικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, φωτομηχανικές, λέει, ε, αντιγραφές. Μπορεί αυτό να, γίνει, να ξεπεραστεί, δηλαδή να ξεπεραστούν οι φωτομηχανικές από ψηφιακές. Το ίδιο ισχύει από τα ιδιωτικά αντίγραφα. Ε, συζητήθηκε στην Γερμανία επί πολύ εάν πρέπει να απαγορευτεί και, η ψηφιακή, και το ψηφιακό ιδιωτικό αντίγραφο Βεβαίω το ψηφιακό ιδιωτικό αντίγραφο δεν μπορεί να ελεγχθεί από το δημιουργό. Πρέπει να επιτρέπεται λοιπόν και στον ψηφιακό τομέα υπό την προπόθεση πάντοτε ότι προσφέρεται στο δημιουργό δίκαιη αντιστάθμιση. Και αυτό όμως προϋποθέτει ένα ευρωπαϊκό δίκαιο προστασίας του δημιουργού και ένα σύστημα νομοθετημένο αντιστάθμισης, αποζημίωσης, το οποίο πρέπει να προβλέπεται σε ενωσιακό επίπεδο. Διότι η ένωμη κατάσταση όπως αυτή ισχύει σήμερα που ρυθμίζεται διακρατικά δεν μπορεί να σταθεί πλέον σε μια αγορά που διέπεται από το διαδίκτυο. Τελειώνοντας να πω λίγα λόγια για το ρυθμιστικό οπλοστάσιο. Λιγότερο δίκαιο είναι καλύτερο, αυτό ισχύει και για την πυκνότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων. Μέχρι τώρα έχουμε 10 ρυθμίσεις, 10 οδηγίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το δίκαιο προστασίας του δημιουργού. Αρχικά ξεκίνησε ανατομέα όπως για την προστασία τραπεζών δεδομένων και τα λογισμικά υπολογιστών και ούτε καθεξής. Μετά, με αυτές όμως, στην ουσία πρόκειται για ένα patchwork με κάποιες επικαλύψεις όπως είπε ένας σοφός άνθρωπος και από ό,τι έχω αντιληφθεί ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίθεται να κάνει μια συνολικότερη ρύθμιση παρά μονάχα βελτιώσεις όπου θεωρεί ότι αυτό απαιτείται. Όμως τέτοιες βελτιώσεις αυτού του patchwork δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με μονομένες αποφάσεις του που εν μέρη υπερβαίνουν τις ε, πολιτικές επιδιώξεις των χωρών μελών και που δεν επιτρέπουν να, να δοθεί μια συνολική λύση. Καλύτερα να υπάρξει μια ενοποίηση του νοσιακού δικαίου. Αυτό μπορεί να γίνει και στα πλαίσια μιας πλήρους εναρμόνισης μέσω μιας οδηγίας. Το καλύτερο θα ήταν όμως να εγκριθεί κανονισμός που να έχει άμεση εφαρμογή σε όλες τις χώρες μέλη. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι ένα βαρύ έργο το οποίο δεν μπορεί ε, να δεν μπορεί να γίνει, να επιτευχθεί μέσα στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Έχουμε, όπως είπα ήδη, ένα μεγάλο ε, patchwork από διάφορες ρυθμίσεις, αλλά η πολιτιστική ποικιλία στην Ευρώπη πρέπει να διατηρηθεί. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ καθηγητά. Και τώρα, όλοι οι ομιλητές ήταν τόσο καλοί και σεβάστηκαν τόσο πολύ το χρόνο τους. Έχουμε περίπου 20 λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις. Ο κύριος Μαρδίνιου Ιππίντου ήταν ο πρώτος που ζήτησε να λάβει το λόγο. Λοιπόν, ας, ας είναι σύντομος παρακαλώ και καταγράφουμε τα ονόματα για τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Μαρίνο Ιππίντου. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Είμαστε στην πραγματικότητα ενώπιον δύο πραγματικότητων. Τα δικαιώματα των ε, δημιουργών δεν αντιστοιχούν στην έννοια του copyright η οποία είναι αγγλοσαξονική. Τα δικαιώματα του δημιουργού έχουν και μια ηθική διάσταση που είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί υπάρχει ανάγκη της προστασίας της ακαιρεότητα και της πατρότητας του έργου. Αυτή η διάσταση λοιπόν της ε, ιδιοκτησίας περισσότερο αφορά το θέμα του copyright, το να αντιγράφει ή όχι κανείς ένα, ένα έργο το βασικό χαρακτηριστικό ενός καλλιτεχνικού ε, έργου είναι κυρίως η απόλαυσή του. Όλη η δημιουργία είναι κάτι που έχει στόχο να δώσει κάτι, να το απολαύσει η κοινωνία. Οποιοςδήποτε δημιουργός θέλει να διαβαστεί ή να ακουστεί το έργο του, να το θαυμάσει ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός ατόμων. Από την άλλη πλευρά γύρω από ένα δημιουργό έχουμε ένα σύνολο από συμφέροντα που είναι κυρίως οικονομικού χαρακτήρα και ιδιωτικού χαρακτήρα που δυσκολεύουν την πρόσβαση στο έργο του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει μια νομοθεσία η οποία επιτρέπει την συλλογική απόλαυση του έργου του καλλιτεχνικού, των συγγραφέων ή των συνθετών, των έργων που λόγω της ε, αξίας τους και της διάστασής τους μπορούν να είναι αγαθά κοινά για όλους τους πολίτες καλλιτεχνική δημιουργία είναι κοινωνική από τη φύση της, κοινωνικοποιημένη. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη υποστήριξη προς τους ε, δημιουργούς με τη δημιουργία φόρων στα, στις συσκευέ που κάνουν πιο εύκολη τη χρησιμοποίηση αυτού του έργου και όχι σε βάρος του δημιουργού. Πρέπει λοιπόν να ξεχωρίσουμε την κατανάλωση ενός έργου από το κοινό από την αντιγραφή για στόχους εμπορίας που δίνει τη δυνατότητα σε κάποιο κέρδος για τους ενδιάμεσους. Εκεί πρέπει να είναι η προτεραιότητα στην ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Θέλω να χαιρετήσω ιδιαίτερα την έκκληση για μια νομοθεσία που βασίζεται στα πραγματικά στοιχεία. Αυτό είναι και ο στόχος της Επιτροπής μας για καλύτερη ρύθμιση και νομοθεσία. Ως εισηγήτρια για την οδηγία Ενφοσόκ θέλω και αυτό να το λάβω υπόψη μου και εγώ χαίρομαι που ο καθηγητής Δήμπος ε, μας έχει δώσει τα στοιχεία για την παρουσίασή του ε, δημόσια και αυτό είναι πολύ θετικό για μας. Επίσης, στο δρόμο για την καλύτερη ρύθμιση ο καθηγητής Στύπα έχει κάνει ορισμένε παρατηρήσεις. Πρέπει το copyright να αντέξει και στο μέλλον. Θα ήθελα να ξέρω από τον κύριο Ντούμπος και τον κύριο Κρέτσμερ αν θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να ανοιχτό πρότυπο στον κατάλογο των εξαιρέσεων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις τεχνολογικές εξελίξεις στο μέλλον. Για τον καθηγητή Κρέτσμερ, εσείς αναφερθήκατε στην ε, κουλτούρα αυτή που στον πολιτιστικό τομέα που δεν υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν άδειε. Τα λεγόμενα μέτρα DRM στον τεχνολογικό κόσμο είχαν μεγάλες επιπτώσεις στις βιβλιοθήκες, στα μουσεία κτλ. για να διατηρηθούν τα ψηφιακά έργα όταν τίθενται στο δημόσιο χώρο. Από την άποψη αυτή το copyright λαμβάνει επαρκώς το ρόλο αυτού του, αυτών των θεσμών πολιτιστικής κληρονομιάς για να διατηρήσουν τα ψηφιακά έργα για το μέλλον και και ποια θα είναι η άποψή σα για το θέμα αυτό και επίση προς τον καθηγητή Ντούπο, Κρότσμαρτ και Στύπα θα ήθελα να σα ρωτήσω ποια είναι η εμπειρία σα με τι λεγόμενες ε, επεκτεταμένες συλλογικές άδειε ECL που έχουν ε, χρησιμοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ορισμένε σκανδιναβικέ χώρε μπορούν αυτέ οι επεκτεταμένε συλλογικέ άδειε να βοηθήσουν να υπάρχει μεγαλύτερη χρήση και εκμετάλλευση των έργων και να υπάρχουν μια ευρύτερη εφαρμογή του ECR στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την εδαφική διαθεσιμότητα των έργων. Και τέλος, τέλος, μήπως μπορείτε να συνιστήσετε τη χρήση αυτών των εργαλείων και να ζητήσετε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει και νομοθετικά βήματα ώστε να μπορέσει το ECL να λειτουργεί καλύτερα στον ψηφιακό ενιαίο χώρο. Thank you. Mrs. Triple. Κυρία Τρίπελ, ευχαριστώ πολύ. Έχω ένα ερώτημα στον κύριο Στύπα και στον κύριο Τρόγκ αν αφήσουμε την εδαφικότητα του copyright και την χάσουμε. Τι θα σημαίνει αυτό για την ε, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές λύσεις που μπορούμε να σκεφτούμε. Η κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, ομιλητές που μοιράστηκαν μαζί μας ε, το όραμά τους για το μέλλον των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Διάφορα μηνύματα ακούσαμε, ότι είναι το πρώτο δηλαδή εισόδημα, πηγή εισοδήματος για τους δημιουργούς, πρόκειται για αμοιβή των δημιουργών. Επίσης είναι ένας τρόπος για να ε, αξιοποιηθεί το, η πολιτιστική κληρονομιά της Υπήρου μας η οποία αντιμετωπίζει νέες καινοτόμες προκλήσεις στην ψηφιακή εποχή και μας ε, θα πρέπει να δουλέψουμε ώστε να διατηρηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην εξασφάλιση της πρόσβασης του κοινού σε περισσότερο πολιτισμό και δημιουργία, αλλά ακριβώς και το συνδυασμό αυτού με τη δίκαιη αμοιβή ε, και τη συντήρηση της ε, δημιουργικής φλέβας της Υπήρου μας. Ε, επίσης, να έρθω στο ερώτημα που ήθελα να θέσω. Άκουσα καλά τι είπε ο κύριος Τρόμ, μεταξύ άλλων που μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα, επέμεινε το οικονομικό βάρος του τομέα των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και το τζίρου και τα νούμερα τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί και που θα ακούσουμε σε ορισμένες εβδομάδες είναι πολύ διαφωτιστικά και πολύτιμα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω ε, με βάση αυτά που είπε. Μήπως μπορούσε να με διευκρινίσει σε αυτό το στάδιο, αν είναι δυνατόν, ποια θα μπορούσε να είναι η πρόταση της ΕΖΑΚ για αντισταθμιστική χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών μηχανιών. Πώς θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε κάποια περισσότερα πράγματα για αυτή την πρόταση που μπορεί να υποβληθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Κάστερ. Τονίστηκε προηγουμένως ότι πρέπει να ξεβρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων διαφόρων εμπλεκομένων και εκπροσώπων συμφερόντων. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτή η ισορροπία δεν μπορεί να εξασφαλιστεί κατά από τις διαδικασίες της αγοράς. Εγώ την εντύπωση ότι η ισορροπία μεταξύ των δημιουργών, των καταναλωτών και αυτών που ε, δημιουργούν προσθέμενη αξία αυτή τη στιγμή κατευθύνεται κυρίως στους τελευταίους. Αυτό είναι αποτέλεσμα των διαδικασιών της αγοράς. Μήπως επομένως θα πρέπει όταν εμείς εστιάζουμε στα θέματα του copyright να εξασφαλίσουμε και την ε, υπεροχή της πολιτικής συναντή της αγοράς και το copyright μήπως θα έπρεπε να έχει σαν πραγματικό στόχο να προστατεύει τους καλλιτεχνικούς δημιουργούς και το εισόδημά τους και το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης των καταναλωτών στην καλλιτεχνική δημιουργία. Uh, thank you, Madame Ευχαριστώ, η κυρία Ροζιέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως υπάρχουν κάποια ουσιαστικά θέματα που ακούσαμε εδώ και τα υπενθυμίσαμε. Ήταν πολύ πλούσια η σημερινή ακρόαση. Πάντως συνένεση αποτελεί να έχετε δίκιο, Πρόεδρε, ότι πρόκειται για ένα δικαίωμα πραγματική ιδιοκτησίας, ιδιοκτησίας βασικά. Οπότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα ωφέλη αυτό του δικαιώματος για τους δικαιούχους του, δηλαδή τους δημιουργούς. Και μέχρι στιγμής, αν, ακόμα και αν επικρίθηκε ο τρόπος με τον οποίο έχει οργανωθεί ο τομέας του πολιτισμού, πάντως μέχρι στιγμής οι ε, δημιουργοί είναι βέβαιοι ότι ασκούν το δικαίωμά τους όχι μόνο σε μια δίκαιη αμοιβή, αλλά και το ηθικό τους δικαίωμα για το έργο του, επί του έργου τους, δηλαδή πώς χρησιμοποιείται, πώς ε, εγγυάται κανείς την αυθεντικότητά του. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει επικριτικά να δούμε αυτή την αλυσίδα νέων αξιών που αναπτύσσεται στο τομέα του πολιτισμού, αλλά που νομίζω είναι πρόδρομος μιας ανακατανομής των αξιών σε πολλούς τομείς, διότι έχουμε πρόσβαση, είναι αλήθεια, σε πολιτιστικά αγαθά δωρεάν ε, και αυτό ε, είναι πολύ εκτεταμένο. Αλλά η δωρεάν διάθεση είναι επιφανειακή, γιατί υπάρχουν μέσα διάθεσης δωρεάν, αλλά υπάρχουν και μέσα διάθεσης με προστιθέμενη αξία που όμως απλώς πάει στους διανομείς που ε, έχουν έτσι μια ελκυστική προσφορά, αλλά μετακινούν τη βάση της εργασίας τους σε άλλους τομείς, ας πούμε συλλογή προσωπικών δεδομένων, διαφήμιση και το ε, πολιτιστικό προϊόν δεν είναι πλέον η καρδιά της ε, επιχείρησής τους, αλλά ε, είναι η βιτρίνα. Πρόκειται για παράπλευρους μάλλον τομείς που προτείνονται. Ε, μπορεί κανείς δηλαδή πια να δημιουργήσει ένα εργαλείο, ένα αντικείμενο και θα μπορούσε κανείς να το χρησιμοποιήσει δωρεάν ε, ε, ο διανομέας του και να φτιάξει προστιθέμενη αξία, να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία με εμπορικές προσφορές σε άλλους τομείς. Το βλέπουμε ας πούμε για την πώληση εκινήτων, αγαθών. Το βλέπουμε με ένα σωρό site που το κάνουν αυτό. Είναι και το παράδειγμα των ε, low cost ε, εταιριών που κερδίζουν από άλλου τομεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την μόνιμη αμοιβή των δημιουργών αλλά και την αμοιβή αυτού που στηρίζει τη δημιουργία. Δηλαδή το πρότυπο των πνευματικών δικαιωμάτων όπως υπάρχει θα πρέπει να εξελιχθεί για να προσαρμοστεί στις νέες πρακτικές, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω επίσης ποιες προτάσεις υπάρχουν για να εξασφαλιστεί τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση της δημιουργίας από όλους αυτούς τους φορείς που αυτή τη στιγμή αποκλείονται. The last question by Mr. Ευχαριστώ. τελευταία ερώτηση από τον κύριο Διακόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οποιαδήποτε συζήτηση, όπως έχει πει, είχε πει ο Βολτέρος, θα ήταν καλό να συνεχίζεται για δύο-τρεις εβδομάδες ή και περισσότερο και να καταλήγει πρώτα σε ορισμούς, γιατί η ίδια η συζήτηση ε, δεν μπορεί να γίνει σύντομα. Και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Στύπερ, ότι πρέπει να ορίσουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Και οι όροι είναι πολύ διαφορετικοί από τη μια χώρα στην άλλη. Έχουμε μια σειρά ε, πολιτιστικών προϊόντων. Ορισμένα είναι εργατέχνη, άλλα είναι αντίγραφα. ή αντιπροσωπεύουν άλλου είδους προϊόντα. Αν μπορούμε λοιπόν να ορίσουμε μια ιεραρχία αυτών των νοημάτων, αυτών των ενιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες, ποσοστά, αμοιβέ, ε, συστήματα για τη συλλογή των αποζημιώσεων μπορεί να και, γίνουν και σε εθνικό επίπεδο είναι η άποψή μου ότι αυτοί οι όροι πρέπει να οριστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκούς ορισμούς και μια ιεραρχία που να υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα υπόλοιπα είναι δευτερευούσε σημασία και μπορούν να γίνουν σε εθνικό επίπεδο. Συμφωνώ με τον κύριο Πίντο και άλλους που ε, μίλησαν για την ηθική συνιστόσα του δικαιώματος του πνευματικού, δηλαδή η κυριότητα του καλλιτέχνη και του έργου, που δεν αναφέρεται μόνο σε χρήμα, αλλά σημαίνει την εγγύηση της ακαιρεότητας του ίδιου του έργου. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Ε, τώρα θα δώσω το λόγο στους ε, καλεσμένους μας για να απαντήσουν. Αν μπορούν όσο γίνεται πιο σύντομα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Είναι δύσκολο για μένα να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μια-δύο. Καταρχήν, νομίζω πως τα συμφέροντα των δημιουργών και των επενδυτών είναι διαφορετικά. το παράδειγμα του ηθικού δικαιώματος που έδωσαν δύο μέλη είναι καλό, γιατί όντως εκεί δεν συμπίπτουν τα <laughs> συμφέροντα. το ηθικό δικαίωμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να διαπραγματευτεί. Δηλαδή, δεν μπορεί να το διαπραγματευτεί ο δημιουργός με τον ε, ε, δικαιούχο της άδειας εκμετάλλευσης. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ο εφευρέτης της ασπιρίνης, ο Φίλιξ Χόφμαν, που έφτιαξε το, την ασπιρίνη το 37, πέθανε το 46. Τα δικαιώματα για την ασπιρίνη τα είχε η Bayer, που ήταν η εταιρεία που εργαζόταν αυτός. Η μεταφορά του δικαιώματος έγινε λόγω της σύμβασης. Αν όμως σκεφτείτε τη δημιουργική συμβολή ενός εφευρέτη που είναι παρόμοια με τη δημιουργική συμβολή ενός, ε, ε, ε, ενός δημιουργού, η ασπιρίνη, πάλι θα πήγαινε στην πάγεν. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι μεγάλες οι προκλήσεις που προκύπτουν από την μεταφορά του δικαιώματος από τον δημιουργό στον εκμεταλλευόμενο το δικαίωμα. Τώρα για την ECL ε, ε δεν έχουν γίνει πολλά ε, για τις, ομαδικέ, για τις εταιρείες διαχείρισης ομαδικά δικαιωμάτων. Νομίζω στις σκανδιναβικές χώρες έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες, μεγάλα προγράμματα ψηφιοποίησης, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα αν έχουν επιτύχει ή όχι. Τώρα, για ανοιχτά, ανοιχτές προδιαγραφές, νομίζω ότι θα ήταν κάτι ωφέλιμο, αλλά και πάλι θα πρέπει να δούμε ποιε ε, είναι οι επιπτώσεις όλων αυτών. Δηλαδή θα πρέπει κανείς να ερευνήσει και αυτό είναι το βασικό μήνυμα που εγώ έχω να σας δώσω, ότι πολλά από αυτά τα θέματα πρέπει να, να ερευνηθούν με εμπειρικό τρόπο. Δεν χρειάζεται να ρυθμιστούν ε, ε, μόνο με συζήτηση. Να απαντήσω μονάχα σε δύο ερωτήματα που αναφέρθηκαν σε μένα για τον κλειστό κατάλογο εξαιρέσεων και το αν υπάρχει ανάγκη να είναι ανοιχτός ο κατάλογος αυτός θα ήθελα να αναφερθώ και στην έκθεση διαβούλευσης. Αυτό το οποίο μπορείτε να δείτε εκεί και το ακούσαμε όλοι σήμερα από τους εμπειρογνώμονες. Πολλοί εκπρόσωποι χρηστών, ομάδες χρηστών και θεσμικοί χρήστες είναι αυτοί οι οποίοι ζήτησαν να υπάρχουν ανοιχτοί κατάλογοι εξαιρέσεων, γιατί υπάρχουν νέες πρακτικές και νέες τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται πλέον. Υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη, όπως παραδείγματος το περιεχόμενο το οποίο δημιουργείται από τους χρήστες. Γι' αυτό οι εμπλεκόμενοι αυτοί θέλουν να υπάρξουν αλλαγές στον κατάλογο των εξαιρέσεων και περιορισμών. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο αναφέρθηκε είναι η, το ECL, οι εκτενείς συλλογικές άδειες. Εδώ έχουμε σημαντικούς ε, θεσμικούς χρήστες οι οποίοι αγωνίζονται και έχουν να αντιμετωπίσουν και τις ρήτρε εδαφικότητας των ε, αδειών. Αυτό αποδείχθηκε πολύ θετικό για να λύσει το πρόβλημα που ανέφερε ο Μάρτιν Κρέτσμερ στην αρχή όταν έδειξε το χάσμα αυτό του 20ου αιώνα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε ψηφιωμένα βιβλία. Με τις συλλογικές άδειε θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό της πρόσβασης σε βιβλία τα οποία δεν είναι πια σε κυκλοφορία. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να δώσει και μια νέα πηγή εισοδήματος για τους καλλιτεχνικούς δημιουργούς, τους συνεγραφείς και θα, δώσει, θα έδινε και μεγαλύτερες δυνατότητε για ευρύτερη πρόσβαση. Θα σας ενθάρρυνα λοιπόν να δείτε μερικές από αυτές τις βέλτιες πρακτικές που υπάρχουν. Είναι το Bocaux πρόγραμμα στην Νορβηγία που έχει ψηφιοποιήσει πάνω από 100.000 βιβλία και προσπαθούν να ψηφιοποιήσουν ό,τι είναι γραμμένο στα νορβηγικά και έχει δημοσιευτεί μέχρι το 2000 αλλά λόγω της εδαφικότητας της ρήτρα ECL θα μπορούν να το χρησιμοποιούν μονάχα χρήστες που έχουν διευθύνσεις IP Νορβηγίας. Μα αυτό δεν είναι κάτι που θέλουμε σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και εγώ να δώσω μια γενική απάντηση στις διάφορες παρατηρήσεις και τα ερωτήματα για τη διαβούλευση σε σχέση με το copyright. Εκπρόσωπο μία από τις ε, μεγαλύτερες οργανώσεις στην Ευρώπη και τις οργανώσεις των συγγραφέων ήμουνα όλοι, ήμασταν όλοι σε πάρα πολύ παράξενη θέση όταν έγινε αυτή η διαβούλευση. Ήταν 80 ερωτήματα τα περισσότερα των οποίων σπρώχνανε τον ε, απαντώντα σε μία κατεύθυνση ή σε κάποια άλλη. Όλα αυτά τα οποία πρέπει να προστατεύσει η Κομισιόν, το Ακή Κομινοτέρο, όλα αυτά ήταν μέσα στα ερωτήματα. Συγχρόνως υπήρχαν κάποια σχέδια που είχαν δημιουργηθεί από κάποιες ε, ομάδες κοινωνικές για να υπάρξει μια απάντηση κατά του copyright. και ορισμένοι λέγανε ακριβώς τα ίδια πράγματα κατά του copyright. Σαν συγγραφέας κανείς θα πρέπει να δει πώς θα προστατεύσει τα δικαιώματα των δημιουργών. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό και εγώ προσπάθησα να σας δείξω με τα στοιχεία και με τα σχόλια που χρειάζεται να υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις και που δεν χρειάζεται να υπάρξει αλλαγή. Γιατί, όπως προσπάθησα να παρουσιάσω, δεν Προσπάθησα να εξηγήσω λοιπόν όλα αυτά. Σε αυτή την άσκηση λοιπόν πολιτική στην Ευρώπη θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έρχονται διάφορα email από πολλέ κατευθύνσει. Δεν ξέρετε από πού προέρχονται όμω. Αν τα μετράτε σαν μεμονωμένε απαντήσει υπάρχει ένα κίνδυνο. Γι' αυτό υπάρχει και ένα μητρό διαφάνεια για να μπορεί κανεί να είναι ε, αξιόπιστο στις απαντήσεις. 11.000 απαντήσεις, ναι. Αλλά εκπροσωπούνται ένα εκατομμύριο δημιουργοί. Μία απάντηση ενός δημιουργού μετριέται σαν μία, ένα, ενώ μια οργάνωση που εκπροσωπεί χιλιάδες δημιουργών θεωρείται και αυτή σαν μια ενω μια απάντηση. Όλο αυτό πρέπει να το δούμε λιγάκι πιο προσεκτικά. Είδαμε κάποια στοιχεία της έρευνας που είναι πολύ χρήσιμη για τους ε, ε, λήπτες αποφάσεων. Αλλά δεν είναι μόνο η έρευνα που έχει γίνει, πρέπει να δείτε και τις άλλες έρευνες που έχουν γίνει. Υπάρχουν και τελεολογικού αριστοτέλειου χαρακτήρα έρευνες. Και κάπου έχουν προαποφασιστεί τα αποτελέσματα και οι, τα στοιχεία συλλέγονται για να επιβεβαιώσουν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά συμφέροντα τα οποία πρέπει να εξορροπηθούν, πρέπει να ακούσετε τις απόψεις όλων αυτών και πρέπει να δείτε πώς η αγορά επηρεάζει τους καταναλωτές στην ευρωπαϊκή οικονομία και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να σταθεί ισχυρότερη αν των τρίτων χωρών και όχι να έχετε μονάχα μία έρευνα που αφορά μία συγκεκριμένη περίπτωση και ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. ο κύριος Στούπερ ότι οι χρήστες, οι καταναλωτές ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για τα θέματα του copyright. Στο παρελθόν απλώς παίρναν τα έργα αυτά από τον, μέσω του εμπορικού τομέα. Τώρα έχουμε τα κοινωνικά μέσα και έχουμε ένα άλλο τρόπο για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά. Οι παραδοσιακές εταιρείες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όταν δεν θέλει κανείς να πληρώσει τα τέλη για τη μουσική, λένε ότι αυτό γίνεται λόγω των καλλιτεχνικών δημιουργών. Ενώ αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν πληρώνουν τους δημιουργούς. Και εδώ έρχομαι στο θέμα αυτό που ανέφερα στο τέλος και εκεί ζήτησε κάποιος περισσότερη πληροφορία. Η μεταφορά αξίας πρέπει να αντιμετωπιστεί προσεκτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές αμοιβή πρέπει να αντιμετωπιστεί ενδεχομένω και από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αλλά πρέπει με τον τρόπο αυτό να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα τα οποία ε, ωφελούνται από το περιεχόμενο θα πρέπει και αυτοί να δίνουν κάποια αμοιβή στους <clears throat> δημιουργούς από τους οποίους προέρχεται ένα έργο. Ευχαριστώ. Να σας πω ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο, λίγα λεπτά μονάχα, διότι έχουμε και κάτι διερμηνήσει εδώ. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ ευγενικό, αλλά σας παρακαλώ είστε σύντομοι. Για να απαντήσω το ερώτημα της κυρίας Τρίπλ. Και σχόλιο. Έχει δίκιο η κυρία Τρίπελ, γιατί οι ε, διατάξεις αποκλειστικότητας και εδαφικότητας είναι εκ των όνων κάνευ στις συμβάσεις για την προχρηματοδότηση οπτικοακουστικών έργων. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Ευχαριστώ. Εγώ για να απαντήσω στις ερωτήσεις έχω δύο σχόλια. Αρχίζω το τέλος. Όπως διαπιστώσατε στην ερώτηση σας αρχικά, όλοι εκπλησόμεθα ότι μεταξύ των 10 προτεραιοτήτων της Ευρώπης περιλαμβάνεται και η περιλαμβάνεται και η ισοπαίδωση του δικαίου του δημιουργού. Νόμιζα ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Βρισκόμαστε στην εποχή της αυθονίας σε όλους τους τομείς. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση, ο κόσμος έχει αλλάξει σε έργα καλλιτεχνικά, μουσικής κτλ. Έχουν τώρα πρόσβαση οι καταναλωτές σε 20-30 εκατομμύρια έργα, κάτι που δεν υπήρχε ποτέ. Τεχνικά μπορεί αυτό να βελτιωθεί, αλλά προς Θεού, ας συγκεντρωθούμε στα πραγματικά διακυβεύματα για τους Ευρωπαίους. Ακόμα και οι πλέον πρόσφατες χρήσεις ε, του διαδικτύου και δυστυχώς εδώ οφείλω να φέρω αντίρρηση σε όλους τους ε, πανεπιστημιακούς εδώ καλύπτονται από άδειε όλα τα περιεχόμενα που, φτιάχνουν, ε, που δημιουργούν οι χρήστες. User generated content. Ας μην εξακολουθούμε να επιμένουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και ας δούμε ξανά ποιες είναι οι προτεραιότητες της Ένωσης. Παρ' όλα αυτά υπάρχει, υπάρχουν μέσα στα μοντέλα της νομοθεσίας και που έχουμε, είναι ο λόγος της αποτελεσματικής αποδοτικότητας μας και των χιλιάδων θέσεων εργασίας. Διότι στην, καταστρέψαμε από την άλλη μεριά όμως την βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη με ατελείς και ημιτελείς ρυθμίσεις. Έχουμε δαπανίσει δισεκατομμύρια των φορολογουμένων, δεν έχουμε ωστόσο τελικά ένα ευρωπαϊκό Google ή άλλο τίποτα σχετικό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ρυθμίσουμε και το τελευταίο πρόβλημα που είναι της ψηφιακής εξαίρεσης που δημιουργήθηκε με την Οδηγία Ηλεκτρονικού Εμπορίου του 2000 και που βάζει φραγμός το δικαίωμα που αναγνώρισε ωστόσο η Οδηγία του 2001. Εμείς αναγνωρίσαμε το δικαίωμα ε, αποζημίωσης των δημιουργών. Δεν υπάρχει λόγος να ξανανοίξει αυτό. Το πρόβλημα είναι η οδηγία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Είτε λοιπόν τώρα θα ξανανοίξετε την οδηγία του ηλεκτρονικού ε, εμπορίου και θα πρέπει να λυθούν πολλά προβλήματα και της ε, προστασίας της προσωπικής σφαίρας και Ευχαριστούμε πολύ. Ζητήσει γνώμη από τους Διερμηνείς διότι τους έχω τρυπεί αυτιά. Είτε θα περιοριστούμε μονάχα στο πρόβλημα των, ε, ε των δικαιωμάτων του δημιουργού, οπότε θα πρέπει να δούμε την αντίφαση μεταξύ της οδηγίας του 2000 και του 2001. Ο νόμος Google, ο γερμανικός νόμος Google, αλλά είναι ο τύπος ο Που που πλουτίζει ε, από τους από τον τύπο. Γιατί, Γιατί κάθε δευτερόλεπτο το Google ρωτάει όλα τα site του κόσμου όπως και τα site του τύπου και λόγω της ποιότητας ε, της παραγωγής των Ευρωπαίων ε, δημοσιογράφων το Google πλουτίζει. Εγώ όταν διαπραγματεύτηκα με το YouTube διαπραγματεύτηκα, αλλά με το Google νομίζω ότι μπορώ να διαπραγματευτώ. Γιατί εξαίρεση ε, ηλεκτρονικό εμπόριο οδηγία του 2000. Δεν είναι ότι δεν συμφωνούν για δίκαιη αμοιβή. Δεν θέλουν καν να συζητήσουν μαζί μας. 96% των εισοδημάτων προέρχονται από τις άδειες. Οπότε η οδηγία του 2000 είναι αυτή η οποία εμποδίζει Πρέπει να αναθεωρηθεί αυτό το σύστημα, να επιβληθεί μια ισότιμη αμοιβή που λαμβάνει υπόψη τον πλούτο που δημιουργείται χάρη στο προστατευμένο ε, πολιτιστικό περιεχόμενο για τους μηχανισμούς έρευνας, τα... για τις μηχανές αναζήτησης στο ίντερνετ, όπως η Google. Ο καθηγητής Τίπερ, ευχαριστώ. Θα έρθω μόνο σε δύο θέματα η κατήσχηση της πολιτικής απέναντι στην αγορά, ε, μίλησε κάποιος. Εγώ βρίσκω επικίνδυνη διατύπωση αυτή απέναντι στο δικαίωμα προστασία του δημιουργού, διότι η προστασία του δημιουργού υποτίθεται ότι δημιουργεί αγορά για το καλλιτεχνικό δημιούργημα. Συνδέοντας απαγορεύσεις ή προσφέροντας απαγορεύσεις στον δημιουργό, δίνουν τη δυνατότητα να χορηγηθούν άδειες Χρειάζεται λοιπόν αυτό για να δημιουργηθεί η αγορά για τις άδειε. Από αυτό συνεπάγεται επίσης ότι μπορώ να περιορίσω το δικαίωμα προστασίας του δημιουργού στη δημιουργία ενός τέτοιου πλαισίου δικαίου για την αδειοδότηση προϊόντων. Δεν χρειάζεται επομένως να ρυθμιστεί περισσότερο η αγορά αυτή και αυτό αναφέρεται και στους φραγμούς που επιβάλλει το δίκαιο προστασίας του δημιουργού απαραίτητο είναι αυτό εκεί όπου δεν μπορεί από μόνη της να λειτουργήσει μια αγορά. Αυτό δεν λαμβάνεται συχνά υπόψη. Υπάρχουν φραγμοί για την χρήση σε περιπτώσεις όπου λειτουργεί ή θα λειτουργούσε το σύστημα της αδειοδότησης, όπου ωστόσο έχουν επιβληθεί φραγμοί που δεν μπορούν ωστόσο να υποκαταστήσουν την λειτουργία της αγοράς. Και γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά την δημιουργία του ανοιχτού φραγμού του λιγόμενου, του λιγόμενου, της λεγόμενης έντιμης χρήσης, η δίκαιης χρήσης που, ε, για την οποία μιλούν οι Ηνωμένε Πολιτείε, που σημαίνει ότι μπορούν να διατηρήσουν οι χώρες μέλη πάλι όλους τους εθνικούς φραγμούς τους, πάλι λοιπόν δεν προκύπτει εναρμόνιση και από την άλλη μεριά μπορεί στο επίπεδο των κρατών μελών με επίκληση αυτής της γενικής ρήτρας να επιτραπούν κάποιες χρήσεις οι οποίες δεν αφαιρούνται από την αγορά διοδοτήσεων. Γι' αυτό είναι καλύτερο να επιτευχθεί μια ευελιξία ανοίγοντας τους φραγμούς να θεσπιστούν δηλαδή στενές γενικές ρήτρες όχι μια πολύ γενική ρήτρα που να λέει επιτρέπεται ότι δεν απαγορεύεται αλλά να είναι σαφές σαφής ο σκοπός της χρήσης. Για παράδειγμα, για παραθέσεις από έργα. Οι παραθέσεις αυτές έχουν ως σκοπό να αποδείξει κανείς ένα επιχείρημα. Εφόσον δεν το χρησιμοποιεί γι' αυτό, δεν είναι απαραίτητο να είναι προστατευμένες. Πρέπει λοιπόν, λοιπόν να είναι συνδεδεμένο με τον σκοπό χρήσεως. Και τελευταίο κάτι το οποίο δεν είπα πριν για λόγους χρόνου. Και βέβαια στο επίπεδο της Ένωσης πρέπει να προστατευτεί και το δικαίωμα του δημιουργού να μην παραμορφώνεται το έργο. Κάτι το οποίο δεν τόλμησαν ακόμα να ρυθμίσουν μέχρι, μέχρι τώρα, διότι και εκεί υπάρχουν πολύ δια, μεγάλες πολιτιστικές διαφορές μεταξύ των χωρών μελών. Είναι όμως κάτι το οποίο θίγει τον πυρήνα τον ίδιο της προστασίας του δημιουργού και το πνεύμα του έργου του δηλαδή, αλλά και την ακαιρεότητά του. Και εκεί απαιτείται εναρμόνιση στο επίπεδο της Ένωσης. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Κάποια τελικά σχόλια για αυτή την ακρόαση. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας και στα μέλη τα οποία έλαβαν το λόγο να σας ε, διαβεβαιώσω, να σας ότι το ενδιαφέρον το οποίο έχει δημιουργηθεί για αυτή την ακρόαση ήταν τεράστιο και ήταν πολύ δύσκολο να αποφασίσουμε ποιος θα προσκληθεί για να λάβει το λόγο σήμερα και σε ποια θέματα, για ποια θέματα. Για αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι ότι δεν εκπροσωπήθηκαν επαρκώς στις συζητήσεις της σημερινής μέρας, λέω το εξής. Ελάτε σε επαφή με τη γραμματεία της Επιτροπής μας και ε, κάντε γνωστές τις απόψεις σας. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε σε κάποια από τις συνεδριάσεις που θα κάνει η ομάδα εργασίας στους επόμενους μήνες. Πρέπει απλώς να ξέρουμε ποιοι είσαστε. Σας παρακαλώ κάντε τους εαυτούς σας γνωστούς σε εμά. Δεν νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτά τα οποία λέγεται σήμερα σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη του copyright στην Ευρώπη. Απλώς θέλω να πω ένα πράγμα. Η ακρόαση αυτή δείχνει, χωρίς καμιά αμφιβολία, ότι το θέμα αυτό βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα για πάρα πολλούς ανθρώπους, μια μορφή ομάδα ανθρώπων, εταιριών, και άλλων εμπλεκομένων. Είτε είναι και απλοί πολίτες οι οποίοι θέλουν να έχουν φτηνή και άμεση πρόσβαση στο καλλιτεχνικό περιεχόμενο, είτε είναι κράτη τα οποία θέλουν να διαφυλάξουν την εθνική ή περιφερειακή τους πολιτιστική ταυτότητα. Είτε πρόκειται για δημιουργούς και μεμονωμένους ερμηνευτές και καλλιτέχνες, οι εταιρείε που ξεκινούν στο ίντερνετ, ή σε μεγάλους ομίλους που θέλουν να έχουν μια απόδοση στο κεφάλαιο που επενδύουν μέσω μιας δίκαιας ανταμοιβή για το, τη χρήση των έργων τους ή για, με αποζημίωση για την παράνομη χρήση. Όλοι αυτοί έχουν λόγο να υποστηρίζουν το copyright. Εμείς ως νομοθέτες έχουμε το καθήκον να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι διεκδικήσεις θα μπορέσουν να εξεταστούν στο νέο περιβάλλον που είναι η ψηφιακή οικονομία και η ψηφιακή κοινωνία. Έχουμε κάνει κάποια μικρά βήματα προς την κατεύθυνση αυτής της τελευταία θητεία του Κοινοβουλίου. Θα αντιμετωπίσουμε τις οδηγίες για τα όρφανα έργα και την διαχείριση συνολικών δικαιωμάτων και την πολυεδαφική αδειοδότηση της μουσικής επιγραμμικά, αλλά δεν τα καταφέραμε τόσο καλά όταν πρόκειται για την ιδιωτική αντιγραφή. Δεν ε, ισχυριζόμαι ότι έχω βρει τις απαντήσεις. <clears throat> Ούτε καν ότι υπάρχουν κάποιες εύκολες απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω παρόλα αυτά ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την πνευματική διαπτυσία και τη μεταρρύθμιση του copyright καθώς και το προσωπικό μας θα χρησιμοποιήσουν όλα τα αναλυτικά στοιχεία που μας δώσατε και τα στοιχεία για καλύτερη ρύθμιση για να εξασφαλίσουμε ότι οι σωστές ερωτήσεις θα τεθούν και ότι η σωστή ισορροπία θα επιτευχθεί όταν πρόκειται για τη μελλοντική πορεία του copyright στην Ευρώπη. Και θέλω να δώσω το λόγο για να κλείσουμε και στην κυρία Κώστα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω μόνο ότι έχω την εντύπωση ότι το πολύ διαφοροποιημένο σενάριο που μας παρουσίασαν οι εμπειρογνώμονές μας, τους οποίους ε, και ευχαριστώ, και από τις ερωτήσεις και από την ολόκληρη συζήτηση βλέπουμε πως ε, αυτή η πρόκληση οφείλεται στην έλλειψη ισορροπία ανάμεσα στου δημιουργού, από την μια πλευρά και την απέτηση δηλαδή προστασίας της δημιουργικότητας και θέλω να θυμίσω και την ε, ε, πολιτιστική και γλωσσική διαφορά που είναι από τα αγαθά που προστατεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από την άλλη πλευρά ε, την απέτηση του χρήστη. Και έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν άλλες μη ισορροπημένες έτσι, ε, προοπτικές. Αν σκεφτούμε την ε, σειρά της ε, την ε, αλυσίδα αξίας της ε, βιομηχανίας της ε, οπτικοκουστικής βλέπουμε ότι έχει πολλά να δει απέναντι στο παγκόσμιο ορίζοντα. Πρέπει λοιπόν να νομοθετήσουμε με ισορροπημένο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη όλες όλα τα συμφέροντα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε η αξία του έργου, το ηθικό και οικονομικό δικαίωμα του δημιουργού να προστατευτεί μέσα στο πλαίσιο των πολυάριθμων νέων εφαρμογών όπου αφορούν την κυκλοφορία των δημιουργιών, των ε, έργων και θέλω να είμαι σαφής σε αυτό γιατί αναφέρθηκε και προηγουμένως Είναι λοιπόν κάπως διαφορετικό το πλαίσιο που εκφράζεται αυτή η νέα εξισορρόπηση που θα δημιουργηθεί και που εξάλλου βλέπει και την απέτηση μιας ε, πιο ανοιχτής ε, οπτικής από πλευράς ε, των ε, καταναλωτών. Θα πρέπει να προσέξουμε και χαίρομαι που αυτό τονίστηκε, πρέπει να προσέξουμε ε, το σενάριο όπου οι μεγάλοι φορείς που δεν είναι Ευρωπαίοι κατά κάποιο τρόπο έχουν συνηθίσει το κοινό και μάλιστα το νεαρό κοινό στην έννοια του δικαιώματος στο δωρεάν πολιτιστικό αγαθό και έτσι υποτιμά και την ηθική αξία του έργου, αλλά επειδή ξέρουμε πως δεν είναι τίποτα δωρεάν, και σε αντάλλαγμα προσφέρει στους διαφημιστές ευκαιρίε οι οποίες δεν είναι καθόλου δωρεάν, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι εδώ πρόκειται για ε, παράκαμψη στην ουσία του δικαιώματος του δημιουργού. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα ισότιμο πεδίο για όλους τους φορείς. Ε, σκέφτομαι την ε, οπτικοκουστική βιομηχανία που έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα και τους φορείς που από ό,τι φαίνεται δημιουργούν ένα περιβάλλον και μια συγκέντρωση και αυτό θα πρέπει επίσης να το πούμε στην Ευρώπη που δεν επιστρέφει την επένδυση και τον και ούτε σέβεται όλους τους κανόνες για την ευρωπαϊκή πολιτιστική δημιουργία, για παράδειγμα, σε σχέση με το μεγάλη χρήση που γίνεται για το, ε, τα πολιτιστικά αγαθά. Εμείς θέλουμε να μπορούν να κυκλοφορούν τα έργα, ενίσχυση της οπτικοακουστικής και πολιτιστικής βιομηχανίας στον ψηφιακό κόσμο και βέβαια να βρούμε και αυτές τις εξαιρέσεις και συμφωνώ με τα όσα είπε πριν ο καθηγητής Τίπερ, ότι δηλαδή μάλλον χρειάζεται να επαληθεύσουμε ποιες θα μπορούσαν να είναι κάποιες ρήτρε οι οποίες ε, να μας βρουν σύμφωνους σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, αλλά και για εκείνους ε, που χρησιμοποιούν τα έργα χωρίς να κερδίζουν, αλλά και αυτούς που κερδίζουν από την, τα δικαιώματα της άδεια εκμετάλλευσης. Όλα αυτά πρέπει λοιπόν να τα εξετάσουμε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ σημαντικά. Είδαμε πόσο πρόκληση, βεβαίως πιστεύω πως η Κομισιό μας θα λάβει υπόψη όλες αυτές, όλους αυτούς τους προβληματισμούς και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την ομάδα εργασίας που έχουμε κοινή, την Επιτροπή Τζούρι και ευχαριστώ ακόμη μια φορά τον Πρόεδρο Σβόμποντα. Πιστεύω πως θα υπάρξουν και άλλε ευκαιρίες στην Επιτροπή μας με τους συνάδελφους της Επιτροπής Πολιτισμού ώστε να εμβαθύνουμε περαιτέρω σε όλες αυτές τις πτυχές. Ευχαριστώ και πρώτου κλείσουμε θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς για τον πρόσθετο χρόνο που μας έδωσαν και κλείνω τη συνεδρία. και οι διερμηνείς ελπίζουν ότι καταλάβατε κάτι από αυτά που ακούσατε αγαπητοί ακροατέ του διαδικτύου.